Welcome to this uh, uh, Καλώς ορίσατε στη συνεδριασή μας. Ξεκινάμε και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε δερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από μαλτέζικα, κροατικά και ιρλανδικά. Αργότερα κατά τη διάρκεια της συναντησής μας θα έχουμε μια ομάδα επισκεπτών από την Εθνοσυνέλευση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας ε, σε επίπεδο πρόεδρων ε, πρόεδροι για παράδειγμα από την ε, νομοθετική επιτροπή συγγνώμη, από την Επιτροπή Νομοθετικής Συμμόρφωσης θα τους καλωσορίσουμε όταν φτάσουν αργότερα Σημείο 3 τώρα της ημερήσιας διάταξης, μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Ε, σημείο 2. Ε, δίνουμε τον λόγο στη Γιώτα να μας κάνει μια ενημέρωση για την επίσκεψη στις αντιπροσωπείας της ΕΜΠΛΑ στη Βόσινγκτον τον Απρίλιο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω για την αποστολή μας που πραγματοποιήθηκε 19 έως 21 Απριλίου 2017. Εγώ ήμουν επικεφαλής ως ε, εκπρόσωπος του Προέδρου της Επιτροπής μας, Τόμας Χέντελ, και στόχος μας ήταν να ε, μιλήσουμε με τους Αμερικανούς εταίρους για ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ε, ε αυτοματοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, ε, νέες εργασιακές σχέσεις και ταυτόχρονα ε, συζητήθηκαν ε, εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης υπό τη νέα κυβέρνηση Τραμπ και τις προθέσεις της στον τομέα της ψηφιοποίησης, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και στο πλαίσιο αυτό συναντηθήκαμε με υπουργεία, με κοινωνικούς εταίρους, με διεθνείς οργανισμούς, με think tank και ιδιαίτερα σημαντικό, ε, σημαντική ήταν η συνάντησή μας με τον καθηγητή Τζόζεφ Στίγκλιτς, τον βραβευμένο με Νόμπελ, ε, καθηγητή πανεπιστημίου. Ήταν πολύ ολοκληρωμένη συζήτηση που ε, διεξάγαμε. Διαπιστώσαμε πολλά κοινά σημεία, ιδίως ως προς την, προς την πρόκληση της ψηφιοποίησης στον ε, στην απασχόληση. Συζητήσαμε ποιες ε, θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν, ποιες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, πώς θα, πώς θα ε, μεταβληθεί η ποιότητα της εργασίας. Διαπιστώσαμε όμως και κάποιες διαφορές μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχουμε διαφορετικά κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, διαφορετικά, διαφορετικές ε, ως προς τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Θα μπορούσα να σας τα λέω για πολλή ώρα γιατί, ε, γιατί ήταν ε, πολύ έντονες αυτές οι τρεις ημέρες της αποστολής. Ωστόσο έχετε στα χέρια σας και την αναλυτική έκθεση που συντάξαμε έπειτα από την επιστολή, την οποία και μπορείτε να συμβουλευτείτε αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος ίσως να προσθέσει κάτι. Όχι, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σα διάταξης. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα ξεκινήσω δίνοντας τον ε, λόγο στην Επιτροπή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τζόρντι Κουρέλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την ε, πρόταση και πιο συγκεκριμένα την εκτίμηση αντικτύπου. Έχω μια παρουσίαση που μπορείτε να δείτε στην οθόνη, οπότε θα ξεκινήσουμε ε, αμέσω. Να σας εξηγήσω στα γρήγορα τι θα καλύψει αυτή η παρουσίαση, μια επισκόπηση της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου. Δεν θα πω στις ιδιαιτερότητες, διότι τις γνωρίζετε. Και μετά θα περάσουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι, στα κύρια απορίσματα της εκτίμησης αντικτύπου σε τέσσερις τομείς ε, επιδόματα ανεργίας, πρόσβασης ε, οικονομικών ενεργών πολιτών σε κοινωνικές παροχές, ε, παροχές μακροχρόνιας φροντίδας και οικογενειακές παροχές. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την εκτίμηση αντικτύπου. Έχουμε ένα συνολογικό βημάτων που βοηθούν τις υπηρεσίες κομισιών και τους συνομοθέτες να διαρθρώσουν την προετοιμασία μιας πρότασης, να έχουν ε, στοιχεία που θα υποστηρίξουν τη χαράξη πολιτικής. Η, η λέξη κλειδί είναι υποστήριξη. Όταν μιλάμε για τέτοια οικονομικά ή κοινωνικά θέματα, τα πράγματα δεν είναι, μαθημα... δεν αριθμητική ένα σε ένα κάνουν δύο. Ε, χρειάζονται πληροφορίες για να γίνεται μια επιλογή βάση πληροφοριών να καλύπτονται μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όλες οι παροχές και όλα τα κόστη και όλες οι επιπτώσεις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα, καλύπτονται όλες οι πρωτοβουλίες από τη χάραξη πολιτικής μέχρι τα μέτρα υλοποίησης. Και μετά, όπως ξέρετε, στην Κομισιόν έχουμε δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή που ελέγχει όλες τις εκτιμήσεις αντικτύπου, ώστε να υπάρχει μια διασφάλιση καλής ε, και ουδέτερης συνεργασίας. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ποιος είναι ο σκοπός της πρότασης αυτής. Ουσιαστικά το να συνεχιστεί ο εξυγχρονισμός ε, των ευρωπαϊκών ε, κανόνων ε, συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μέσω τεσσάρων τρόπων. Όταν κινείται ένας πολίτης από τη μια χώρα στην άλλη, εξασκεί το, ασκεί το δικαίωμα ελευθερής κυκλοφορίας, αλλά αν κάποιος που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάσει τις κοινωνικές του παροχές, ακόμη και δεν τον εμπόδισε κανείς να ασκήσει το δικαίωμα σε κριτικότητα, το έχασε. Οπότε μέσω του εξυγχρονισμού θέλουμε να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος, να διασφαλίσουμε νομική σαφήνεια, δίκαιη και ισότιμη κατανομή του οικονομικού βάρους μεταξύ των κρατών μελών και πρόθεση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ε, διοικητικής απλούστευσης και σωστή εφαρμογή των κανόνων. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα και το πρώτο που μπορείτε να μας προσάψετε είναι ότι η εκτίμηση αντικτύπου είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατική, αλλά επειδή καλύπτουμε τόσους πολλούς τομείς, ήταν δύσκολο να είναι μικρότερη. Επίσης παρέχουμε μια περιλήψη σε όλες τις γλώσσες της πρότασης και έχουμε δημοσιοποιήσει τη θετική γνωμοδότηση αυτής της Επιτροπής, του Internal Board ε, της ε, Επιτροπής που ανέφερα προηγουμένως. Η μέθοδος εκτίμησης που περιλαμβάνει τρία στάδια πρώτα απ' όλα ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε σχέση με μια γραμμή βάση η οποία είναι υπάρχουσα κατάσταση. Μετά υπάρχει ανάλυση των άλλων επιπτώσεων, περιπτώσει απάτης, κατάχρησης, ρυθμιστικών χρεών, δίκαιης, δίκαιο καταμερισμού των βαρών. Και τρίτον, γίνεται μια συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Και εδώ έχουμε δύο επίπεδα ανάλυσης Εδώ βλέπετε τις πηγές που χρησιμοποίησαμε, είναι πολύ επίκυλες. Ε, ε, υπάρχουν δημοσκοπήσεις ε, πανευρωπαϊκές, όπως για παράδειγμα για το εργατικό δυναμικό, η έκθεση για τη γύρανση, τα σύνορα δεδομένο της Eurostat. Της Eurostat. Επίσης, στον τομέα αυτό της κοινωνικής ασφάλισης, ε, σκοπός είναι ο συντονισμός. Ε, περισσότερο οπότε συνεργαστήκαμε στενά με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της Διοικητικής Επιτροπής για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, δεν προέρχονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από εθνικές πηγές. Και επίσης, ε, πέραν από τους ειδικού που μιλήσαμε στην Κομισιόν, να συζητήσαμε και με ειδικού από την Deloitte, την Fresco Network, ε, την ε, HIVA, ένα δίκτυο πολύ ωφέλιμο. Στο πλαίσιο της εκτίμησης που έγιναν και διάφορες διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονε απο από κράτη-μέλη εδώ και περίπου δύο χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της Διοικητικής Επιτροπής κάναμε μια συνάντηση με τους Κοινωνικού εταίρου τον Ιούνιο του 2015 και με τη ΜΚΙΟ τον ίδιο μήνα και είχαμε και δύο δημοσίες διαβουλεύσεις online το 2013 και το 2015. Θα ξεκινήσω τώρα με την πύρινα της πρότασης. Ε, η πρώτη πτυχή αφορά τις παροχές ανεργίας, ε, τα επιδόματα ανεργίας. Κάποιος που ζητά δουλειά σήμερα μπορεί να λάβει επίδομα και να το εξάγει σε ένα άλλο κράτο για περίοδο τριών μηνών με πιθανή επέκταση στους έξι. Σκοπός είναι ο αναζητών εργασία να μπορέσει να βρει μια δουλειά σε ένα άλλο κράτο ε, και να έχει κάποια προστασία. Οι υπηρεσίε απασχόληση τη ε, αρχικής του χώρας, ε, της χώρας καταγωγής του, μπορεί να ζητήσουν μια έκθεση των δραστηριοτήτων του, ετούντος, ε, του αναζητούντος εργασία από την χώρα φιλοξενίας. Μια μηνιαία έκθεση. Εδώ έχουμε κάποια νούμερα. Βλέπουμε ότι στο βασικό σενάριο 27.000 άνεργοι έχουν εξάγει τα επιδόματα ανεργίας τους το 2013-2014. Αντιστοιχεί αυτό μόλις το 0,1% του εργαζόμενου πληθυσμού. Εξετάσαμε διάφορες επιλογές ε, που βλέπετε στον πίνακα αυτών. Έχουμε το βασικό σενάριο, το σημερινό ουσιαστικά, ως πρώτη επιλογή. Μετά έχουμε επιλογή ένα, το να παραταθεί η περίοδος εξαγωγής των επιδομάτων από τους 3 στους 6 μήνες. Ε, αυτή είναι η βασική αλλαγή που εξετάζεται από αυτή την επιλογή. Και μετά το να διατηρηθεί φυσικά ανοιχτή το ενδεχόμενο τέτοιες επέκταση. Και η δεύτερη επιλογή είναι να επεκταθεί η εξαγωγή του επιδόματος αυτού για όλη τη διάρκεια ε, του δικαιώματος αυτού. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη επιλογή είναι να προταθεί η επέκταση παράταση αυτής της περίοδου εξαγωγής από τους 3 στους 6 μήνες. Αυτό βλέπουμε και στην πρόταση που έχουμε υποβάλει. Η δεύτερη πτυχή που σχετίζεται με τα επιδόματα ενεργείας ε, είναι με αυτό που ονομάζουμε aggregation, συρροή. Ε, e. Είναι ένας τεχνικός όρος, πολύ σημαντικός. Ε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άνεργος έχει εργαστεί σε πολλά κράτη-μέλη μπορεί να ζητήσει να λαμβάνονται κατά συρροή e υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης στα άλλα κράτη-μέλη ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο καλύπτει την περίοδο που απαιτείται για να έχει δικαίωμα για επίδομα ενεργεία. Για παράδειγμα, εάν στη χώρα Α, για να έχει κανεί δικαίωμα για επίδομα ενεργεία, πρέπει να έχει εργαστεί για 24 μήνε, απλά το επινοώ τώρα. Αν κάποιο λοιπόν δούλεψε σε ένα άλλο κράτο μέλο για 18 μήνε και μετά έρθει σε αυτό το νέο κράτο μέλο και εργαστεί και εκεί για 8 μήνε, για να εκτιμηθεί κατά πόσο έχει δικαίωμα για επίδομα ενεργεία, δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι οκτώ μόνο τελευταίοι μήνες ε, εργασίας στην τελευταία χώρα. Θα ληφθούν υπόψη και οι 18 μήνες κατά τους οποίους εργάστηκε σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό ονομάζεται συρροή. Όπως έχει σήμερα η κατάσταση, οι κανόνες δεν καθορίζουν ελάχιστο διάστημα προηγούμενης απασχόλησης στην ε, κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο εργάστηκε για 25 μήνε σε ένα κράτο μέλο και μετά πάει σε ένα νέο κράτο μέλο και διαργαστεί και για μία μέρα, θα έχει δικαίωμα για επίδομα ανεργία ε, όπω ισχύει στο νέο κράτο μέλο. Αυτό δημιουργήσε κάποια προβλήματα, οπότε το εξετάζουμε. Να σας δώσω κάποια νούμερα για αυτό. Έχουμε περιπτώσει ροή στην Ευρώπη, ανθρώπων δηλαδή που μετακινήθηκαν και ζήτησαν τέτοια ροή ε, μιλάμε για 25.000 σχεδόν περιπτώσεις, ε, το 41% των οποίων ε, είχαν εργαστεί για λιγότερους από τρει μήνες στο νέο κράτος μέλος. Έχουμε εξετάσει διάφορα σενάρια. Η πρώτη επιλογή ήταν η επισημοποίηση αυτού που έχουμε σήμερα, δηλαδή ότι η συρροή αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά την πρώτη μέρα εργασίας. Η δεύτερη επιλογή θα ήταν να εισηχθεί μια ελάχιστη περίοδος ε, ασφάλισης ενός μήνα στο νέο κράτος μέλος και η τελευταία επιλογή θα ήταν η εισαγωγή αυτής της ελάχιστης περίοδου ασφάλισης αλλά μέχρι τρεις μήνες. Αλλά να είναι τριών μηνών. Ε, αποτιμήσαμε τις δυνατότητες αυτές και κατέληξαμε στο συμπέρασμα όπως ε, αναφέρουμε και στην πρότασή μας ότι η καλύτερη επιλογή είναι να εισαχθεί ελάχιστη, απέτσι ελάχιστη διαστήματος ασφάλισης τριών μηνών. Αυτό κάναμε για τα θέματα συρροής. Και τέλος, και πάλι όσον αφορά τα επιδόματα ενέργεια, έχουμε το ζήτημα των διασυνοριακών εργαζομένων. Σήμερα λοιπόν η κατάσταση έχει ω εξή. Ένα άνεργο διασυνοριακό εργαζόμενο πρέπει να ζητήσει επίδομα ενέργεια στο κράτο μέλο όπου κατοικεί. Και το κόστος των επιδομάτων ενεργείας ε, ε, καταβάλλεται από το κράτος μέλος όπου εργάστηκε, όπου ε, ε, έκανε ασφαλιστικές εισφορές ε, για ε, τους τελευταίους πέντε μήνες. Και εδώ έχουμε κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία, οι διασυνοριακά εργαζόμενοι είναι, πλησιάζουν περίπου τους 800.000 και αυτοί που έχουν εργαστεί για πάνω από 12 μήνες ε, είναι σχεδόν 1,6 εκατομμύρια. Εξετάζουμε λοιπόν και εκεί τις διάφορες επιλογές και καταλήξαμε σε έξι επιλογέ. Η πρώτη είναι ότι ο διασυναρικός εργαζόμενος αποφασίζει ο ίδιο πού θα ζητήσει το επίδομα ενεργεία. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι το κράτο τη τελευταία δραστηριότητα θα πληρώσει το επίδομα ενέργεια και ο... εκεί πρέπει να εγγραφεί ο διασυνοριακός εργαζόμενο. Διότι ξέρετε, σε κάποια κράτη-μέλη η συνθήκη να πάρει κανεί το επίδομα ενεργεία δεν είναι μόνο το πόσο καιρό έχει απασχοληθεί, αλλά το ότι πρέπει ενεργά να αναζητούν εργασία κάποιο Και υπάρχει αυτή η συνθήκη της εγγραφής. Μετά έχουμε την επιλογή 3, η περίπτωση αυτή που επιλέξαμε, την πρόταση το κράτος της τελευταίας δραστηριότητας να καταβάλει το επίδομα ενεργείας μόνο μετά από επαρκές διαστήμα εργασίας, μόνο δηλαδή για παράδειγμα μετά από 12 μήνες εργασίας στο εν λόγω μέλος, τότε θα έχει την ευθύνη το κράτος μέλος εργασίας να καταβάλει το επίδομα ανεργίας. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα στο άλλο κεφάλαιο, την πρόσβαση των οικονομικά ενεργών πολιτών στα κοινωνικέ παροχές. Θα σας το πω συνοπτικά για να περάσω το χρόνο, κωδικοποιήσαμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, πολλές ε, ε, Υποθέσει ε, όπου αποφασίστηκε ότι υπό του κοινού κανόνε υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση στα κοινωνικά ωφέλη από οικονομικά ανένεργου πολίτε. Και αυτό που κάναμε ουσιαστικά είναι ότι κωδικοποίησαμε την ομολογία του δικαστηρίου. Οπότε θα περάσω αυτό το κομμάτι. Τώρα πάμε στο ε, πρώτο κεφάλαιο που είναι οι παροχέ μακροχρόνια φροντίδα. Όπω έχουν τα πράγματα σήμερα παρατηρούμε αύξηση των παροχών στον τομέα αυτών διότι όπως γνωρίζουμε γυράσκουν οι κοινωνίες μας και χρειάζονται όλο και περισσότερα οι άνθρωποι λόγω αυτού. Αυτές οι παροχές δεν ε, αναφέρονται εδώ στον, σε κάποιο κανονισμό και ε, παρέχονται ως παροχές ε, ασθενείας. Οπότε θέλουμε ένα νέο κεφάλαιο όπου θα καθορίζονται οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας και θα αντιμετωπίζονται όπως και σήμερα ως παροχές ασθενείας. Οπότε δεν έχουμε αλλαγή στην πρόταση. Η μόνη αλλαγή στην πρόταση είναι ε, ε, η επεξήγηση όπως κάναμε για τους οικονομικά ενεργούς ε, πολίτες. Ουσιαστικά κωδικοποιήσαμε τις πρακτικές που υπάρχουν. Πάμε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο τα οικογενειακές παροχές. Το πρώτο που βλέπουμε εδώ είναι ότι δεν έχουμε προτείνει αναπροσαρμογή και προτείνουμε επικυροποίηση των κανόνων ε, για τα ε, επιδόματα ανατροφής παιδιού. Θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα αυτό του κάθε γονέα ξεχωριστά και τα κράτη-μέλη θα έχουν την επιλογή να τα πληρώσουν εξ ολοκλήρου και στους δύο εργαζόμενους γονείς. Αυτό σύμφωνα με τη, σημερινή, με τη, με τη μορφή της κοινωνίας σήμερα. Κοιτάξαμε το υπαρκτό σενάριο, το βασικό σενάριο που έχουμε σήμερα βάσει στοιχείων από τα 17 κράτη-μέλη και έχουν δαπανηθεί σημαντικά πόσα σε οικογενειακές παροχές, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Αντιστοιχεί όμως αυτό σε κάτω από το 1% των συνολικών δαπανών σε οικογενειακά επιδόματα, σε μετρητά στις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως βλέπετε κάποια νούμερα που λέμε είναι υψηλά, αλλά αν τα συγκρίνει κανείς με τις συνολικές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τόσο υψηλά. Οπότε τι κάναμε, είδαμε τις διάφορες προτάσεις Και όπως κοιτάμε την αναπροσαρμογή, είχαμε δύο δυνατότητες, ε, είτε προσαρμογή στα στάδια διαβίωσης ε, ε, προς τα πάνω και προς τα κάτω ή μόνο προς τα κάτω. Θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται την αριθμική αναπροσαρμογή. τώρα όσον αφορά αυτό το δεύτερο κομμάτι της πρότασης, έχουμε προβλέψει διάφορους κανόνες ε, συντονισμού ε, των ε, επιδομάτων. Το ένα σχετίζεται με το μισθό, το άλλο ισχύει με υποχρεωτικά επιδόματα και με προαιρετικά επιδόματα. Προτείνουμε διάφορες αλλαγές ώστε να ευθυγραμμιστεί η κατάσταση με τις κοινωνίες μας όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και σε άλλες περιπτώσεις το μόνο που κάναμε είναι ότι διευκρινίσαμε τους κανόνες ώστε να είναι πιο εύκολη στην εφαρμογή. Σταματά εδώ. Ζητώ συγγνώμη που μίλησα τόσο γρήγορα και ζητώ συγγνώμη που η ομιλία μου τρίξε πάνω από 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το, το λόγο στην κυρία Γρίβα από το EPRS για να μας κάνει την παρουσίαση της. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε τα όσα έχουμε κάνει και θα σας εξηγήσω καταρχήν η μονάδα για την ε, προληπτική αξιολόγηση επιπτώσεων, πώς ετοιμάζεται και θα σας πω τι εντοπίσαμε εμείς ε, ως βασικά να σας πω πως έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για το κείμενο αυτό, το οποίο είναι πάνω από 2.000 σελίδες και νομίζω ότι είναι η πιο πλήρης ψηφιολογική μελέτη που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Καταρχήν να σας πω πως το βασικό σώμα της εργασίας μας είναι η αξιολόγηση των επιτοσιολογικών μελετών που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν νομοθετείται κάποιο κείμενο και βέβαια η στήριξη των ε, επιτροπών του Κοινοβουλίου με επιπλέον ε, πτωσιολογικές μελέτες, έτσι ώστε οι επιτροπές σας να μπορούν να πετύχουν τους στόχους της καλύτερης νομοθέτησης και των ε, τεκμηριωμένων αποφάσεων, έτσι ώστε να μπορείτε κι εσείς να ελέγχετε καλύτερα το εκτελεστικό σας όργανο. Να σας πω πως καταρχήν ε, απευθυνόμαστε στις ε, ε, επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν τον κυρίαρχο λόγο σε κάθε γνωμοδότηση και βλέπουμε πως εγώ αυτό που κάνω είναι στέλνω ένα σημείωμα, ένα briefing με τα βασικά στοιχεία της επιτουσιολογική μελέτης όπου αναλύουμε μεθοδολογικά ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά, κάτι το οποίο ετοιμάζουμε εσωτερικά στη μονάδα μας. Να τονίσω πως εμείς επί της ουσίας της πρότασης δεν κάνουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό που αξιολογούμε είναι την ποιότητα της επιτουσιολογικής μελέτης και κατά πόσο σέβεται τους κανόνες περί αυτής που έχουμε στους κατευθυντήρες γραμμές του 2015 για την καλύτερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί τη βάση της απόφασης των συντονιστών, οι επιτροπές σας μπορούν να μας ζητήσουν παραπάνω δουλειά, δηλαδή μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επιπτωσιολογικής μελέτης αυτής, των τροπολογιών, της ουσίας, του σώματος κτλ. Υπάρχουν τρόπος, Υπάρχουν τρόποι ε, για να ζητήσετε κάτι τέτοιο και αυτό βρίσκεται στο εγχειρίδιο ε, που ε, ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2013 η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Και αυτά πάντα στα πλαίσια της προσπάθειας για καλύτερη νομοθεσία. Να σας πω πώς ακριβώς αξιολογούμε την επιτουσιολογική μελέτη. Καταρχήν, αρχικά, προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε μια εύκολη εισαγωγή στο υπόβαθρο και στο σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας και να αξιολογήσουμε πώς η επιπτωσιολογική μελέτη αντιμετώπισε τα επτά ερωτήματα στα οποία καλείται οποιαδήποτε επιπτωσιολογική μελέτη να απαντήσει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό. Ποιες είναι οι επτά ερωτήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η κλίμακα του προβλήματος. Γιατί θα πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι ποιοι είναι οι στόχοι Ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ποιοι είναι οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιοντολογικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτική ε, ε, λύσης, πώ συγκρίνονται μεταξύ τους και ποιες είναι οι διευθετήσει για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Και συνήθως έχουμε τη συνεκτικότητα και συνέπεια της, ε, της γενικότερης μεθοδολογίας για παράδειγμα. Υπάρχει λογική συνέπεια στην επιχειρηματολογία που έχουν προταθεί και αποκρίνονται σε επτά ερωτήσει στις οποίε αναφέρθηκα. Επίσης, ε, σχέση κόστου κόστου-οφέλου και ε, συνέπειε και αποτελέσματο. Επίση, αξιολογούμε την ποιότητα των δεδομένων, όπω επίση και την έρευνα η οποία έχει ε, λάβει η χώρα πριν προετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ψυχολογική Μελέτη κατά πόσο όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορεί έχουν ερωτηθεί ε, καταλήλως. Έχουμε τη 12, ε, την περίοδο των 12 εβδομάδων που πρέπει να τρέξει. Επίσης, τι γίνεται με το Regulatory Scrutiny Board δηλαδή το κανονιστικό επιπτικό συμβούλιο, συμβούλιο που θα πρέπει ε, να δει το κείμενο και επίσης αν έχει χαρτογραφηθεί η ε, πρόταση καταλήλους και αν έχει μελετηθεί ε, η επίπτωσή της με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Και θέλουμε με αντικειμενικό τρόπο να αξιολογήσουμε κατά πόσο τα τεκμήρια που έχουν συμπεριληφθεί είναι χρήσιμα και σωστά έτσι ώστε να αξιολογήσετε εσείς την πρόταση. Όμως, όπως είπα και δεν ε, αμφισβητούμε την πολιτική ε, σκοπιά από την οποία ε, κατευθύνεται μια πρόταση. Και να σας πω ότι κοιτάμε κατά πόσο έχουμε θετικά και αρνητικά, δηλαδή πως εδώ για παράδειγμα είναι τα μακροπρόθεσμα επιδόματα, τα κοινωνικά επιδόματα για όσους δεν είναι δραστήριοι, τα επιδόματα ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόματα. Και εδώ νομίζω ότι αποτελούμε ένα ρόλο που μας επιτρέπει να πούμε πως πρόκειται για μια ε, σφραγιλή πρόταση που κάνει κάποια ερωτηματικά και στα θετικά θα πούμε πως εντοπίζει τα αντίστοιχα προβλήματα σε όλους από αυτούς τους τέσσερις τομείς και ε, εξηγεί ε, τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Επίσης αναφέρεται με τον κατάλληλο τρόπο στην ελεύθερη μετακίνηση ατόμων και τεκμηριώνει πως ε, ο κίνδυνος για τουρισμό επιδομάτων, για προνοιακό τουρισμό, είναι μικρός. Επίσης, αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για να κατανοήσουμε καλύτερα ποια είναι αυτά. Δηλαδή, η έλλειψη διαφάνειας, νομικής βεβαιότητας για τους πολίτες και για τους θεσμούς, μη ίση μεταχείριση για τους πολίτες που είναι σε αντίστοιχη θέση, όπως επίσης και μια έλλειψη ισορροπίας στην κατανομή του οικονομικού βάρους. Τελικά καταλήγουμε πως οι εναλλακτικέ επιλογές που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το αντιμετωπίσει είναι αρκετές και για τα τέσσερα και πρέπει να σας πω πως στην επιπτωσιολογική μελέτη δίνουμε δύο επιπλέον εναλλακτικέ προτάσεις σε σχέση με τη βασική οπότε ε, αξιολογούμε 33 ε, εναλλακτικέ. δηλαδή λέμε ε, κανονιστικό, οικονομικό και κοινωνικό κομμάτι της επίπτωσης σύμφωνα με το βασικό σενάριο έτσι όπως μας λέει η νομοθεσία για την απλούστευση και τη βελτίωση των νομοθυμάτων. Και λέμε, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε θετική ή καμία ε, επίπτωση σε κοινωνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, σε όλα εκτός από τα επιδόματα ανεργίας για τους ε, ε εργαζόμενους τρίτης κατηγορίας που θα οδηγούσε σε μια αύξηση στην κατηγορία αυτή της τάξης του 6%. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αναλύουμε όλες τις επιπτώσεις κάθε εναλλακτικού σενάριου, δηλαδή κανονιστικό, απάτη, κατάχρηση, δίκαιη κατανομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και οι προτινόμενες έχουν ένα κανονιστικό κόστο το οποίο έχουμε κρίνει ασήμαντο ή, επουσιώδος. ασήμαντο ή Και πρέπει να σας πω ότι βασίζεται σε μια σειρά από ε, σφαιρικές εξωτερικές έξι που για το συντονισμό των οικογενειακών ε, επιδομάτων και τη μείωση των ε, επιδομάτων ανεργίας στηρίζουν την Κομισιόν και τρεις άλλες μελέτες έχουν να κάνουν με τη μακροπρόθεσμη περίθαλψη και τα επιδόματα ανεργίας. Χρησιμοποίησαμε επίσης και κάποιες μελέτες από ένα δίκτυο ανεξάρτητων ε, μελετητών στο θέμα της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2015. Η Κομισιόν είπε ανοιχτά πως ε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμού στα δεδομένα που έχει και στα σενάρια βάσης και αρκετά, και αρκετά τους οι οποίοι ε, ε, συζήτησαν τα θέματα αυτά έδωσαν τη γνώμη τους στην, ε, σε δύο φάσεις. Μία το 2013 για τα μακροπρόθεσμα επιδόματα ανεργίας και το συντονισμό αυτών και μία το 2015 ε, που έγινε για τα επιδόματα ανεργίας και, και το συντονισμό των οικογενειακών επιδομάτων. Και πρέπει να σας πω πως για τα συστήματα ε, κοινωνικής ασφάλισης κάναμε και μία ε, ακρόαση τον Ιούνιο του 2015 και άλλη μία ε, επαφή τον Οκτώβριο του 2015. Το 2015 ήρθαμε και σε επαφή με μη καπαόμικρον γνωμοδότηση και η διαβούλευση στα κράτη-μέλη έγινε με εντελεχή τρόπο και μέσω της Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και μέσω ε, δύο ε ε, ε, ε, διαδικασιών διαβουλεύσεων που έγιναν διαδικτυακά. Τώρα, τα αρνητικά. Παρόλο που έγινε αυτή η ευρεία διαβούλευση, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή οι εμπλεκόμενοι δεν είναι έτοιμοι να στηρίξουν κάθε μία από τις ε, δυνατότητες. Και για τα συστήματα και το συντονισμό αυτών, ε, για κάποια κράτη-μέλη έχουμε πιο πολλά στοιχεία από ό,τι για κάποια άλλη. Για παράδειγμα, για την οριζόντια εναλλακτική ε, εναλλακτικό σενάριο για το βασικό δεν έχουμε επαρκή ε, συντονισμό και έχουμε και, την, ε, το σενάριο 3 που είναι τα ε, επιδόματα ενεργεια για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους. Εκεί έχουμε την ίδια δυναμία και βεβαίως αυτό και συμβαίνει και στην περίπτωση των επιδομάτων τέκνων και όλα αυτά τα εντοπίσαμε μετά από σχόλια των κρατών μελών στην διοικητική ε, Επιτροπή και βέβαια η Κομισιόν το εξέφρασε με απόλυτη διαφάνεια. Τα κράτη-μέλη, ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν γνωμοδοτήσει με περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι κάποια άλλα και τα έχουμε διαβουλευτεί περισσότερο. Και δεδομένου ότι η Διοικητική Επιτροπή για το συντονισμό των κοινωνικών, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει ε, συντάξει κάποιε εναλλακτικέ λύσεις και έχει δώσει πληροφορίες για αυτές, καλό θα ήταν για την εργασία που έχει κάνει να μα έχει δώσει πιο πολλέ πληροφορίε, οι οποίε να είναι διαθέσιμε και δημόσια. Πάντως, από τις συναντήσεις του 2016 ε, προκύπτει πως πάρα πολλά καινούργια στοιχεία έχουν αναρτηθεί τώρα στο διαδικτυατικό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο εντοπίσαμε είναι πως η σύνδεση μεταξύ αυτής της πρότασης και της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων δεν έχει ε, διαπιστωθεί αρκετά, με αρκετή σαφήνεια στην επιπτωσιολογική μελέτη. Γιατί κάποιες τροπολογίες ε, συντονισμού, κυρίως για τους υποαπόσπαση εργαζομένους, είναι της, ε, του πεδίου εφαρμογή αυτής τη επιπτωσιολογική μελέτης, γιατί είναι τέτοια τεχνική του φύση. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η δυνάμη διασύνδεση, πιστεύουμε πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε στο σημείο αυτό να έχει προσφέρει περισσότερε πληροφορίε, όπω είπε και ο κύριος Κορέλο, παρόλο που ακολούθησε πολύ ε, αυστηρή προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εξαιρετικά ε, μεγάλο το έγγραφο, δεν είναι εύκολο να διαβαστεί. το βασικό κείμενο είναι 180 σελίδες, το οποίο είναι πολύ παραπάνω από τις 30-40 σελίδες που έχουμε στις συστάσεις και 46 ε, παραρτήματα, ε, άρα λοιπόν έχουμε πάνω από 2.000 σελίδες, ε, με συγχωρείτε 26 παραρτήματα. Και να σας πω πως ο συμπέρασμα αποτελεί μια καλή βάση έτσι ώστε να αλλάξουμε το τρέχον πλαίσιο συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και έχει εντάξει σε μεγάλο βαθμό τα σχόλια που έγιναν από ε, τη δεύτερη γνωμοδότηση του κανονιστικού συμβουλίου. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζονται περαιτέρω προσοχή, όπως είπαμε το γεγονός πως οι εμπλεκόμενοι θα μπορούσαν να έχουν στηρίξει με πιο διάφορο τρόπο όλες τις εναλλακτικέ λύσεις και να γίνεται και πιο σαφής η σύνδεση με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων που εδώ δεν εμφανίζεται παρκώς. Και τέλος, και, η εργασία της Σχετικής Επιτροπής για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα έπρεπε να είναι πιο διάφανη. Για πιο, λεπτομέ, ε, πιο πολλές λεπτομέρειες, εάν θέλετε, μπορείτε να δείτε και τις αρχικές μας ε, εκτιμήσεις που έχουν και κάποια παρετέρω στοιχεία που ενδεχομένως θα βρείτε ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. For, ε, ε, Ευχαριστούμε για αυτήν την πολύ ολοκληρωμένη εισαγωγή στο θέμα. Θα περάσουμε τώρα στον εισηγητή. Ελπίζω να είναι εδώ. Και τους σκιώδεις. Δύο λεπτά ο καθής. Θα ξεκινήσουμε με, τον κύριο Μπάλας. Παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δυσκολεύτηκα να έρθω στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί. για τόσα, είπε η κυρία που παρουσίασε την εκτίμηση δικτύπου. Έχω δύο ερωτήσει αυτή τη στιγμή, ώστε να μην με γρηγορήσω. Ε, η πρώτη έχει ως εξή. Φαίνεται ότι το 55% των ανέργων βρίσκουν δουλειά μετά από 12 μήνες έρευνα και το 75% μετά από 24 μήνες, όπως προκύπτει από αυτό που δείξατε. Όσον αφορά λοιπόν τις εξαγωγές των δικαιωμάτων ε, για επίδομα ανεργίας, αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα περνάμε, λέμε να περάσουμε από τους τρεις στους έξι μήνες, ε, κάτι που αποτελεί πρόοδο ε, βάσει αυτού που προτείνει η Κομισιόν. Αλλά η ερώτησή μου είναι, είναι αρκετό, δεν θα έπρεπε να ε, χορηγούμε το σύνολο των δικαιωμάτων σε επίδομα ενεργείας για το οποίο έχει συνεισφέρει κάποιος εργαζόμενος όταν βλέπουμε ότι οι άνεργοι κατά 55% βρίσκουν δουλειά μετά από 12 μήνες και το 75% μετά από 24 μήνες. Οπότε δεν είναι πρόβλημα αυτό το εξάμεινο διότι χρειάζεται να γίνεται όλο και μεγαλύτερος έλεγχος σήμερα στους ανέργους ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, ε αναζητούν ε, ενεργά μια δουλειά. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε την άποψη των ανθρώπων που έκαναν την μελέτη αντικτύπου. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την απόσπαση. Εγώ βρεθήκα στην Πολωνία με την συνάδελφο την κυρία Στίβεν την Δευτέρα. Συζητήσαμε για το ζήτημα της απόσπαση, το έντυπο 1, α1 κτλ. Εκεί που υπάρχει ισχυρή σύγκληση, όπως διαφαίνεται, είναι ότι σήμερα πρέπει να εξυγχρονίσουμε το πληροφοριακό σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα, το ESSE, e, που είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγή που δεν είναι ακόμα επαρκή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ψηφιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα ε, επί αυτής της πλατφόρμας ή να καταλήξουμε να φτιάξουμε και μια κάρτα ψηφιακή ε, που να περιλαμβάνει και τα στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης και του δικαιώματος ε, για επίδομα Αυτό δεν θα πρέπει να το βαθύνουμε σήμερα, να το ψάξουμε κάπως περισσότερο. Ευχαριστώ κύριο Σούλτσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που λάβαμε σήμερα έχω πολλά ερωτήματα. Πρώτον, η Κομισιόν με τη μελέτη αντικτύπου της θέλει να ακολουθήσει μια διαδικασία νομοθέτησης βάση στοιχείων και να στηριχθεί σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Ταυτόχρονα όμως διαβάζουμε ότι πολλές φορές αυτά τα αριθμητικά στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα και γι' αυτόν τον λόγο έγιναν συνεντεύξεις με υπαλλήλους από την Υπουργεία των Κρατών Μελών ε, καθώς και άλλα στοιχεία. Ε, πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε αυτές τις, ε, αυτά τα στοιχεία και όταν σε περιπτώσεις όπου δεν καταφέρατε να βρείτε αυτά τα στοιχεία, πώς αλλάξατε τις μεθόδους αξιολόγησής σας. Δεύτερον, συζητήσατε ή μάλλον σας διέθεσαν στοιχεία μόνο 17 κράτη-μέλη. Παραπάνω είναι τα μέλη της, ε, της Ένωσης. Γιατί δεν ε, κατέστη δυνατό να βρείτε στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη. Ίσως τα αποτελέσματα στα οποία θα είχατε καταλήξει να ήταν διαφορετικά. Τρίτον, γιατί δεν επιλέχθηκε ε, η δυνατότητα εξέτασης αναπροσαρμογής, αναπροσαρμογής των επιδομάτων παιδιού Αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά παράγοντας που οδήγησε την όλη διαδικασία της Κομισιόν ήταν απλά και μόνο τα χρήματα. Τέλος. Τι ακριβώς ορίζεται ως οικογενειακή παροχή. Διότι κάθε κράτος μέλος ορίζει αυτόν τον όρο διαφορετικά. Πώς ακριβώς θα μεταχειριστεί η Κομισιόν τα νέα οικογενειακά επιδόματα τα οποία θα εξαρτώνται από το εισόδημα της κάθε οικογένειας. Ευχαριστώ η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση της ε, μελέτη αντικτύπου για το συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Τα ε, έγγραφα... Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διερμηνία, μας ενημερώνουν. Is er nu vertaling naar het Περιμένουμε να δούμε αν λειτουργεί η διερμηνία στα αγγλικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξαναρχίζει η ομιλήτρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πολύ ενδιαφέρουσα και ολοκληρωμένη παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με αυτή την πρόταση για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Έχω να θέσω στην Κομισιόν ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Τα έγγραφα Α1 που είναι προϊόν απάτης κυκλοφορούν ευρύτατα. Αν κάποιος, κάποιο κράτος μέλος λοιπόν έχει να κάνει με ένα τέτοιο έγγραφο που είναι προϊόν απάτης, είναι πολύ λίγα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δεν μπορεί απλά να αγνοήσει το έγγραφο, ακόμη και αν η απάτη είναι προφανής. Πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία, έναν διάλογο, ε, κάτι το οποίο είναι και αναποτελεσματικό διαδικασία και που οδηγεί και σε μεγάλη δυσαρέσκεια στα κράτη-μέλη. Μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει κράτη-μέλη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η απάτη πρέπει να καταπολεμάται. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν στην διάθεσή τους μέσα για την αντιμετώπιση της ε, απάτης και να εξασφαλίζουν την ισχύ και την εγκυρότητα των εγγράφων Α1 που κυκλοφορούν. Γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν πώς ακριβώς ορίζει τελικά την ε, απάτη. Επίσης, είμαι υπέρ του να αυξηθεί ε, ο χρόνος αναμονής στους τρεις μήνες προτού αρχίσει η καταβολή των επιδομάτων ε, ανεργίας. Είναι σημαντικό αυτό ακριβώς για να εξασφαλιστεί ε, μια πραγματική κινητικότητα των εργαζομένων και γι' αυτόν τον λόγο είμαι ε, κατά των, ε, της επέκτασης του χρονικού αυτού περιθωρίου από τους 3 στους 6 μήνες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος καλωσορίζει την ομάδα των επισκεπτών από την Ιγυρία. We have a discussion right now on the Θέλω να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια συζήτηση για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αγαπητοί επισκέπτες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό. Ο λόγος στην κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να θέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Μας υπόθηκε ότι εξετάζοντας το σενάριο βάσης έναντι των άλλων επιλεκτικών, για παράδειγμα τη μη τη αριθμική αναπροσαρμογή των επιδοματών ε, παιδιού και σε συγκρίση με τις συνολικές κοινωνικέ δαπάνες, ότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ρωτήσω ποια είναι η επίπτωση μιας τέτοιας ε, ρύθμισης στους ε, προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Έχετε στοιχεία, αν όχι, γιατί όχι. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Μας υπόθηκε ότι ε, κοιτάζοντας την μελέτη αντικτύπου ότι δεν είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έτοιμοι για όλες τις εναλλακτικές επιλογές. Μήπως όμως πρόκειται για τον εμπλεκόμενο φορέα που είχε την μικρότερη συμμετοχή και συμβολή στην όλη διαδικασία της διαβούλευσης. Τρίτον, είπατε ότι δεν είναι σαφής η διασύνδεση με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Τι λείπει λοιπόν, κατά τη γνώμη σας. Και τέλος, συμφωνώ με τον εισηγητή που είπε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ατομική κάρτα κοινωνικής ασφάλισης για την καταπολέμηση της απάτης. Να επαναφέρω λοιπόν αυτό το ζήτημα της ηλεκτρονικής κάρτας εδώ, που νομίζω ότι θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο να εξεταστεί ως ενδεχόμενο και στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκάμπη Τσίμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την μελέτη αντικτύπου της, αλλά και για την ενημέρωση ε, και τις, εξε... και τις εξηγήσεις που λάβαμε από την υπηρεσία έρευνας του Κοινοβουλίου. Το πρώτο μου ερώτημα σχετίζεται με τις αντιδράσεις και την αξιολόγησή τους. Πρώτον, τα ασφαλιστικά ταμεία στη Γερμανία εκφράζουν τον φόβο τους ότι η θέσπιση ενός αυτόνομου κεφαλαίου για τις ε, παροχές φροντίδας ενδέχεται να αυξήσει τόσο το κόστος συνολικά όσο και να δυσκολέψει την πρόσβαση των πολιτών σε τέτοιου είδους ε, παροχές. Ποια είναι η γνώμη σας. Δεύτερον, η υπηρεσία έρευνας διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας δεν πλήττονται από την πρόταση, ωστόσο επισημαίνει ότι η γαλλική γερουσία θεωρεί ότι ε, παραβιάζονται, παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας. Το εξετάσατε, ποια είναι η δική σας γνώμη. Τρίτον, μιλώ, θα ήθελα να μιλήσω για, την, ε, για τον αποκλεισμό ε, ανίκανων προσεργασία πολιτών τρίτων χωρών. Πώς ακριβώς θα πρέπει να εξασφαλίζεται Πώς ακριβώς πιστεύετε, ε, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στους ε, πολύ φτωχούς ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένετε αύξηση των αστέγων. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους Ρωμά. Ο κύριος εισηγητής αμφισβητεί και την προθεσμία των έξι μηνών. Το ίδιο και εγώ. Ε, εξετάσατε τι είδους και αν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, τι μορφή θα έχουν αν ε, τεθεί σε ισχύ αυτή η διάταξη ε, ε που αναφέρει ότι ε, η καταβολή του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ολόκληρο το χρονικό διάστημα και όχι μόνο τους έξι μήνες. Ευχαριστούμε Τζιν Λάμπερτ. Ήθελα να κάνω δύο σχόλια βάσει και τόσο όσων είπαν οι συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου και τα σχόλια των ενδιαφερομένων, υπήρξαν σχόλια για αυτό το θέμα του πεδίου εφαρμογή, ειδικότερα όσον αφορά τους οικονομικά ανενεργούς, διότι παρατηρούμε μια μεταβολή από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό που βλέπουμε τώρα στη συζήτηση όσον αφορά των ε, δικαιωμάτων Ευρωπαίων υπηκών ε, διασυνοριακά, το βλέπουμε τώρα και με τον Brexit και αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα. Υπάρχει η αίσθηση ότι ορισμένε αποφάσει του δικαστηρίου αντί να γίνονται δεκτέ, θα έπρεπε να είχαν αποτελέσει το αντικείμενο προσφυγής και να εφαρμοστούν τελικά διαφορετικοί κανόνε. Γιατί δεδομένου ότι βλέπουμε πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει ε, προσωρινές δυσκολίες, να ε, ε, επαναπατρίζεται στη χώρα καταγωγής του ή να άνθρωποι και προσωπικό να αντιμετωπίζουν πρόβλημα πιθανής απέλασης. Μήπως πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα έπρεπε οι αποφάσεις αυτές του δικαστηρίου να τις δούμε λίγο πιο επιφυλακτικά, να δούμε λοιπόν αν έχουν ληφθεί σχόλια για αυτές τις αποφάσεις. Έχω μία ερώτηση για τις υπηρεσίες εδώ του Κοινοβουλίου. Συζητάτε για τα κράτη-μέλη και τι ρόλο θα παίξουν, αλλά έλειπαν καθόλου ενδιαφερόμενοι από τις απαντήσεις άνθρωποι που θεωρείται ότι θα έπρεπε να πούν την άποψή τους και να ακουστούν ή μήπως απλά το θέμα αυτό θεωρείται ελάχιστα τεχνικό οπότε, ε, πολυτεχνικό οπότε δεν απαντάνε Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι από του οποίου θα έπρεπε να είχαμε ακούσει κάποια γνώμη, αλλά δεν ακούσαμε. Και όσον αφορά τα νούμερα, ε, τα κράτη-μέλη, αυτό υπήρξε ζήτημα από τότε που ασχολούμαι εγώ με το ζήτημα αυτό, δηλαδή 18 χρόνια και πιθανώ και περισσότερο. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν απαραίτητα ακριβή νούμερα, οπότε αυτό που βλέπουμε εδώ με την αναθεώρηση Μπορεί να συνεπάγεται ότι χρειάζεται να δούμε λίγο και τον κανονισμό για τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πιο σταθερή βάση στο μέλλον. Αντί να παραπονιόμαστε διαρκώ για την έλλειψη στατιστικών στοιχείων κάθε φορά που το κοιτάμε. Ίσως να υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι για του οποίου τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν τα στοιχεία αυτά, ίσως γιατί δεν του βοηθούν να υπερασπιστούν ε, την επιχειρηματολογία τους, οτιδήποτε προσπαθούν να επιτύχουν. Οπότε καλό θα ήταν ίσως να τα δούμε αυτά. Ε, να υπάρξει κάποιος τρόπος στα κράτη-μέλη να υποχρεούνται να δώσουν αυτές τις πληροφορίες ε, τακτικά. Ευχαριστούμε. Η Λαώρα Ατζέ δεν είναι εδώ. Ζωέλ Μελά, θέλετε να πείτε κάτι. Κύριε Μάιτον, έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία της Ζωέλ ε, Μελά, έχει πάει σε επίσημη αποστολή στη Μόσχα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν για την εκτίμηση αντικτύπου καθώς και την ERPS για την πρώτη αξιολόγηση. Τα έγγραφα αυτά, παρότι υπάρχουν και άλλες προφορίες φυσικά, είναι πλήρη και μας διαφωτίζουν όσον αφορά τα διακυβεύματα ε, που συνεπάγεται αυτό ο συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Thank you. Then I'll give the floor to Ο κύριος Μπέκερ λοιπόν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί ήταν μια πραγματικά πολύ επαγγελματική συλλογή πληροφοριών και νομίζω πως ε, η επιπτωσιολογική μελέτη συμπεριλαμβάνει τα όσα χρειαζόμαστε. Θα ήθελα να προσθέσω στα όσα είπε ο Σκιώδης Κάνοντας και τις δικές μου παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τις οικογενειακά επιδόματα και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα επιδόματα τέκνου και το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας πω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πως δεν χρειάζεται να κάνουμε μια προσαρμογή στα οικογενειακά επιδόματα και η δική μου ερώτηση είναι για ποιο λόγο. Γιατί αν δούμε τι γίνεται στις διάφορες περιπτώσεις, νομίζω ότι η αξιολόγηση μας οδηγεί στο αντίθετο συμπέρασμα. Επίσης, αρκετές α, ε, αντιπροσωπείες αναφέρθηκαν στο θέμα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία αποτελούν μια εξαιρετική βάση, ε, από της οποίας μπορούμε να υπολογίσουμε και ένα σωρό άλλα θέματα, για παράδειγμα το μισθολογικό ντάμπινγκ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια επίθεση ε, στα επίπεδα της κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας στην Ευρώπη, πιστεύω ότι αυτό θα ήταν αρνητικό για όλους τους ε, πολίτες μας. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επίτροπη, έχετε τέτοιου είδους σχέδια, ξέρετε να υπάρχουν τέτοιου είδους προθέσεις για μειώσεις. Ο κύριος Λέναρς και ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τα δικά μου σχόλια στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Τώρα για τα επιδόματα τέκνων. Να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσέξει γιατί μας λέει είναι το 1% μη σας ανησυχεί. Ναι, αλλά είναι το 1% είναι και το ποσοστό των ανθρώπων που είναι σε απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν εκεί γιατί είναι αρκετό για να λάβουμε δράση και εδώ όχι. Και μία από τι εναλλακτικέ λύσει που θα πρέπει να δούμε είναι τι θα γινόταν και αν θα ήταν νόμιμο να δώσουμε στα κράτη-μέλη την ευελιξία είτε να επιλέξουν την α, αναπροσαρμογή των επιδομάτων τέκνων, είτε όχι. Το έχετε κοιτάξει αυτό επίσης. Εξαίρεση για τους 3 με έξι μήνες ε, και το επίδομα ανεργίας, πιστεύω, πως είναι ωραία ιδέα να υπάρχει αυτή η εξαίρεση έτσι ώστε να μπορεί κανείς να βρει δουλειά σε αυτό το διάστημα. Αλλά αυτό που ακούω από τους ανθρώπους ε, είναι πως ε, τέτοιου είδους ε, συστήματα πέφτουν θύματα κατάχρησης πολύ συχνά. Και μίλησα με τους βέλους υπευθύνου από τις αρχές και μας είπαν ότι στο Βέλγιο υπάρχει εξή παράδοση. Ο κόσμος θα χρησιμοποιήσει αυτά τα επιδόματα ανεργίας κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού και κυρίως στις χώρες Μεσογείου. Άρα λοιπόν η τάξη που έχουμε ενδεχομένως ε, δεν είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου κατάχρηση θερινοδιακοπών. Ε, θα ήθελα να σα πω λοιπόν πω η επιτουσιολογική μελέτη που μας παρουσιάζεται είναι πάρα πολύ γενικόλογη και θα ήθελα να μα κάνει μία έρευνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δει από πιο κοντά τι σημαίνει όλο αυτό το οποίο παρουσιάζει για τον απλό κόσμο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι από τις κάτω χώρε ε, από μια περιοχή μου πολύ κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Οι κάτω χώρε προσφέρουν ε, ε, επιδόματα τα οποία δεν είναι χρηματικά αλλά είναι σε είδος ε, και το Βέλγιο προσφέρει σε χρήματα αλλά όχι σε είδος. Οπότε, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος που ζει στο Βέλγιο και έχει ε, ε, σύνταξη στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, την ιατρική ασφάλιση την παίρνει από το Βέλιο ε, και στο μέλλον θα παίρνει το κομμάτι των ε, προνοιακών επιδομάτων από την Ολλανδία. Ενώ σήμερα και αυτά προσφέρονται από το Βέλγιο. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει μια ανισορροπία σε επίπεδο καταβολών. Έχει κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο θα επηρεάσει κάτι αντίστοιχο, γιατί πρέπει να το δούμε. Πρέπει να δούμε το θέμα της μακροπρόθεσμης περίθαλψης και Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να οδηγήσει στο να μειωθούν τα προνοιακά επιδόματα που και τα δικαιώματα ανθρώπων που ζουν σε περιοχές γύρω από τα σύνορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν δίνοντα το λόγο στον κύριο Κορέλ για να μας απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα ερωτήματα που πράγματι ευθυγραμμίζονται και με το πνεύμα θα έλεγα της ε, μελέτης αντικτύπου και του προτινούμενου κανονισμού. Πράγματι, σκοπός αυτού του εκτενούς εγγράφου που έχουμε υποβάλει είναι να γίνει μία συζήτηση βάσει στοιχείων. Και φυσικά κάθε πλευρά θα ε, βγάλει τα δικά της ε, συμπεράσματα. Όσον αφορά την εγκυρότητα των δεδομένων. Θέλω να πω ότι αφενός ήμασταν πολύ ειλικρινείς, διότι αναγνωρίζουμε τον, ε, τον περιορισμένο χαρακτήρα των δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα μπορούσαμε και να το είχαμε κρύψει, αλλά θεωρήσαμε ότι στο πλαίσιο της διαφάνειας θα ήταν ορθότερο να αναγνωρίσουμε τα, ε, τους περιορισμούς και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι τα δεδομένα ε, στα οποία στηριχτήκαμε ήταν πολύ χρήσιμα για, για παράδειγμα για τους οικονομικά ανενεργούς ε, πολίτες ε, χρησιμοποιήσαμε στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται ενδεχομένω 100% στον ορισμό του κανονισμού, παρόλα αυτά είναι χρήσιμα και αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, να πω ότι είναι σημαντικό να λάβει κάνει υπόψη του, υπόψη του ότι έχουμε έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν στοιχεία δεν αμφισβητούνται τα στοιχεία αυτά γιατί προέρχονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι εξαντλήσαμε όλες τις δυνατότητες και όλα τα στοιχεία. Εν τούτης, θεωρώ ότι είχαμε ένα επαρκές σύνολο δεδομένων πάνω στα οποία στηριστήκαμε. Για το 1% θέλω να πω ε, ότι πρέπει να έχουμε κατά νου δύο πράγματα. Πρώτον, τους απόλυτους αριθμούς που είναι πολύ ψηλοί σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά πρέπει κανείς να έχει υπόψη του και το ειδικό βάρος ε, αυτού του αριθμού. Όπως είπα, δεν μιλούμε για μια απλή μαθηματική, ε, απλό μαθηματικό τύπο. Ε, έχουμε δεδομένα βάσει των οποίων υποβάλλουμε τις προτάσεις πολιτικής μας. Το άλλο θέμα που τέθηκε αφορά τα επιδόματα ανεργίας. Δύο είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν. Αν θα πρέπει να επεκταθεί η περίοδος ή και αν αυτό ε, αλλάζει την κατάσταση ιδίω όσον αφορά την φροντίδα υγείας. Όσον αφορά την πρώτη πρόταση, είναι ακαθόδες αυτό το ζήτημα. Τα περισσότερα επιδόματα ανεργίας απαιτούν να ε, έχει κανείς ε, συλλέξει δικαιώματα. Δηλαδή συγκεκριμένα να έχεις δουλέψει για κάποια χρόνια και συνέχεια έχεις δικαίωμα να πάρεις ανεργία. Αν αρρωστήσεις δηλαδή, ε, όπως και, και σε περίπτωση που ε, αρρωστήσεις έχεις δικαίωμα να νοσηλευτείς και να λάβεις ιατρική περίθαλψη. Αλλά τα επιδόματα ενεργείας πολλές φορές προϋποθέτουν ότι κανείς θα πρέπει να έχει ενεργά αναζητήσει εργασία. Αυτό απαιτεί όχι μόνο έλεγχο αλλά και υποστήριξη από τις υπηρεσίες εξέβρισης εργασίας στις διάφορες χώρες. Να επεκτείνουμε λοιπόν την περίοδο της εξαγωγικότητας των εξι μηνών θα έδινε, θεωρήσαμε, περισσότερες δυνατότητες στους αναζητούντες εργασίας να βρουν εργασία δηλαδή στο νέο κράτος μέλος, ταυτόχρονα όμως ε, θα υπήρχε και μια απώλεια της επικοινωνίας ε, με τους ανθρώπους αυτούς. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν ότι ε, τα μέτρα ενεργοποίησης θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Για το ζήτημα της απόσπασης, της απάτης και το πώς διασυνδέονται αυτά τα δύο. Είναι σαφές. Υπάρχει σχέση. Το έχουμε δει και σε άλλα θέματα, το έχουμε δει και στη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται σε πολλά κράτη-μέλη σχετικά με τη διοικητική συνεργασία ε, στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων. Αυτό που προτείνουμε εδώ είναι η σαφής βελτίωση της συνεργασίας. Πρέπει να πω ότι η εντύπωσή μας είναι ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι καλή. Τηρείται δηλαδή αυτή η αρχή της καλής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρχών. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις όπου το πράγμα δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά και εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που προτείνουμε Λοιπόν, ιδίω όσον αφορά την απόσπαση, είναι η ενίσχυση των εργαλείων και των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ε, ε, η εφαρμογή των κανόνων και ότι οι εθνικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των αποσπασμένων εργαζομένων. Υπάρχει για το σκοπό αυτό και ο διάλογος μεταξύ των διοικητικών αρχών. Αυτό που είδαμε κατά τις συζητήσεις μας με τους διάφορους εμπληκόμενους φορείς είναι ότι επί της αρχής συμφωνούν όλοι ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες ε, αλλά όταν συζητούμε σε μεγαλύτερο βάθος τι ακριβώς πρέπει να γίνει, εκεί τα πράγματα περιπλέκονται. Ε, Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχει μια καλή βάση προκειμένου Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία για την βελτίωση της συνεργασία. Απάτη εδώ είναι ένα ζήτημα θεμελιώδες. Δεν αφορά μόνο την απόσπαση εργαζομένων. Μιλάμε για ανθρώπους που ενδεχομένω να λαμβάνουν ε, επιδόματα ανεργίας χωρί να, να τα δικαιούνται. Και εδώ έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές που επίσης ενισχύουν την περιοδική ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος ε, ε, των δικαιωμάτων επιδόματος ανεργίας. Το άλλο ζήτημα με το οποίο ε, ασχοληθήκαμε ήταν οι οικογενειακές παροχές και συγκεκριμένα η τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Και εδώ εξετάσαμε και αυτή την πιθανότητα. Δεν την απορρίψαμε εξ αρχής, άλλωστε την εξετάσαμε και στο πλαίσιο της μελέτης αντικτύπους και ε, φτάσαμε στο συμπέρασμα, στο, στη μελέτη αντικτύπου, βάσει του οποίου ε, υποβάλλουμε και τις συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής μας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν πάρα πάρα πολύ επιβαρυντική. Θα ήταν πολύ δύσκολο δηλαδή να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία θα λάμβανε υπόψη όλα τα στοιχεία και όλους τους παράγοντες που θα πρέπει να σταθμίζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή θα καταλήξει σε κάτι που θα είναι δίκαιο. Δεύτερον, οι διοικήσεις, οι διοικητικές αρχές ε, δεν λέω ότι αυτό θα ήταν καλό ή κακό, απλά ε, είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο, θα επιβαρύνονταν πάρα πολύ. Σήμερα η δικτική αρχή που ε, χορηγεί ε, τα, τις οικογενειακές παροχές κοιτάζει την εθνική νομοθεσία και πληρώνει. Αν όμως είχαμε να κάνουμε μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή ε, και ε, έχουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει οικογένεια για παράδειγμα που το, έχει το ένα παιδί στη Σουηδία και το άλλο στη Ρουμανία και ενδεχομένως ο γονέας να ζει είτε στη μία είτε στην άλλη χώρα η καταβολή αυτών των οικογενειακών παροχών ε, θα, θα έπρεπε να περιλαμβάνει τρεις υπολογισμούς. Θα ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Αυτό βλέπουμε είναι αντικειμενικό. Βάσει αυτού λοιπόν βγάλαμε ένα σαφές συμπέρασμα πολιτικής. Η πρόταση αφορά την απόσπαση, ε, τηρεί την αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία, το έχουμε συζητήσει και αυτό εσωτερικά και στον τομέα της τιμαριθμητικής αναπροσαρμογής η Κομισιόν κατέληξε στο ότι θα πρέπει να ε, τηρηθεί η αρχή των ίσων επιδημάτων για ίσα δικαιώματα. Άρα, ε, πρέπει κανείς να έχει ε, ε, πληρώσει στο σύστημα προκειμένου να μπορεί να, βάλει, ε, να, να λάβει επιδόματα. Θα πρέπει να το ζητήσουν κοινοβούλιο και κοινοβούλιο για να καταλήξουν σε συμφωνία. Υπήρξε και ένα ερώτημα για τα εθνικά στοιχεία, κυρία Χάρκιν νομίζω το έθεσε, για το αν έχουμε εθνικά δεδομένα στη διάθεσή μας. Έχουμε, ναι, και μπορώ να σας, να σας τα δώσω αν θέλετε. Ε, για την τιμαριθμική ανα, ανα, ε, ε, αναπροσαρμογή ε, να σας πω ότι η Ιρλανδία πλήρωσε 11 εκατομμύρια σε οικογενικές παροχές στο εξωτερικό. 0,36% των συνολικών δαπανών αυτών. Ε, η τριμαριθμική αναπροσαρμογή θα τροποποιούσε προς τα κάτω βέβαια την, την, την, την πληρωμή των ε, επιδομάτων. Επίσης, τέθηκε το θέμα σχετικά με τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες. Δύο ήταν οι κατηγορίες ερωτήσεων. Πρώτον, αν μειώνουμε τα δικαιώματα και αν αυτό θα έχει επιπτώσεις στην αύξηση των αστέγων κτλ. Εμείς ε, μιλούμε μόνο για τους ε, ε, πολίτες που κάνουν χρήση του δικαιώματος σε ελεύθερης κυκλοφορίας. Ε, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε για την, με την εναρμόνιση σε επίπεδο εθνικού, ε, σε επίπεδο κράτους μέλους. Κάθε κράτος μέλος μπορεί πλέον να αποφασίζει ε, ποια θα είναι τα επιδόματα που θα λαμβάνουν οι πολίτες που κατοικούν στην επικράτειά τους. Αυτό που κάνουμε είναι απλά κωδικοποιούμε τους κανόνες. Φυσικά, ε, η κυρία Λάμπερς έχει δίκιο ότι η νομολογία πολλές φορές μπορεί και να αναιρεθεί. Ε, ως Κομισιόν όμως θεωρήσαμε ότι βασικότερος ε, στόχος είναι να καταπολεμηθεί η απάτη και ο κανονισμός ε, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να, να μετακινούνται από χώρα σε χώρα και ορισμένες φορές ε, έχουμε αυτό το φαινόμενο του τουρισμού των επιδομάτων. Υπάρχουν διάφορες απόψεις επί του θέματος αυτού βεβαίως. Η γνώμη της Κομισιόν είναι σαφής. Για τα μακροχρόνια ε, επιδόματα παροχής εμείς ούτε διευρύνουμε ούτε περιορίζουμε το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας. Ε, κάθε χώρα θα εξακολουθήσει να μπορεί να αποφασίζει μόνη της τους κανόνες, ωστόσο θέλουμε να είμαστε σαφείς, χωρίς να αλλάζουμε την ουσία των ε, κανόνων, ε, ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες που θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν. Αυτά. Θα συνεχίσουμε βέβαια στις συζητήσεις μαζί σας και σε ε, τη συζήτηση μαζί σας σε βάθος για αυτή την πρόταση, όπου και θα έχουμε τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε διάφορα θέματα που μένουν ανοιχτά. Δύο μικρά ερωτήματα. Καταρχήν να ξεκινήσει η κυρία Ρέγνερ, μετά ο κύριο Σούλς και μετά θα το δώσουμε το μικρόφωνο στην στο κέντρο ερευνών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε δυνατότητα το θέσω και εγώ ένα ερώτημα. Στον, ε, στο θέμα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση, φυσικά μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα τη κάρτα ασφαλισμένου. Και εδώ θέλω να πω ότι είπατε κι εσεί ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ καλή. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας εργοδοτών και εργαζομένων από τον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι μας εξήγησαν τι ακριβώς δεν λειτουργεί στον τομέα των εγγράφων Α1. Σε περιπτώσει, για παράδειγμα, που υπάρχουν ε, εργατικά τυχήματα και ε, που ε, μεταφέρεται κάποιο εργαζόμενο στο νοσοκομείο, διαπιστώνεται πολύ συχνά ότι τα στοιχεία που είχε δώσει δεν ήταν σωστά. Γι' αυτό και οι ίδιοι οι εργαδότε ε, απευθύνθηκαν σε εμά λέγοντας ότι ανταγωνιστές τους ε, παρατυπούν και παραβιάζουν τους κανόνες. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις Βεβαίω και στα άλλα θέματα. Είπατε, αναφερθήκατε και στι οικογενειακέ παροχέ και στα επιδόματα τέκνου. Θέλω να σα θέσω το ερώτημα. Τα στοιχεία των εγγράφων Α1, ο έλεγχος, η καλύτερη διασύνδεση και η, η διαπίστωση ότι όλα αυτά λειτουργούν πολύ καλά στην πράξη. Ε, όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καθορίσουν και τα μέτρα που θα αποφασίσουμε να θεσπίσουμε. Κύριε Σούλτσε, συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο, θύμωσα λίγο όμως με το ζήτημα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Ξέρετε ότι δεν συνηθίζω να ξαναπαίρνω το λόγο. Είπατε ότι έχουμε μία μεγάλη συζήτηση εδώ. Και εγώ ακόμη δεν έχω ξεκάθαρη ε, εικόνα. Αυτό που δεν δέχομαι είναι όμως να μου λέτε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα, είναι πολύ δύσκολα. Αν θέλετε να επιτύχετε συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα στην πράξη, πρέπει να εγκαταλείψετε επιτέλους αυτή την τακτική σας, να φέρνετε αυτά τα ακραία παραδείγματα περί οικογένειας, που οι γονεί μένουν σε μία χώρα και το ένα παιδί μένει στην άλλη και το άλλο παιδί στην παράλληλη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να, βασιζό, να βασιζόμαστε σε τέτοιου είδους ακραία παραδείγματα όταν κάνουμε ε, συζητήσεις πολιτικής. Παρακαλώ να εμένετε ε, σε πιο πραγματικά στοιχεία όταν ε, δίνετε τις απαντήσεις σας. Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κορέλ. Είναι πολύ σαφέ το μήνυμα και το λάβαμε. Θα ήθελα να προσπαθήσω να το επαναλάβω. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η επιπτωσιολογική μελέτη και αν είτε μας αρέσει είτε όχι, νομίζω ότι αποδεικνύει πως υπάρχει ένα αυξημένο διοικητικό βάρος για τις αρχές. Ίσως δεν το είπαμε αρκετή σαφήνεια. Ξέρω πως η Επίτροπος κυρία Τάισεν είναι πολύ σαφής ε, στο σημείο αυτό. Εντάξει, αυτό μας λένε τα στοιχεία και η πραγματικότητα αποδεικνύει πως πρόκειται για πολιτική απόφαση η οποία μπορεί να σας βρίσκει σύμφωνος ή όχι. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως επειδή προτείναμε ε, ίσες αμοιβέ για ίση εργασία θα πρέπει να ξεκινάμε επίσης με ίσα δικαιώματα προνοιακά για ίσες εισφορές. Αυτή είναι η όλη προσπάθεια που κάνουμε την επιπτωσιολογική μελέτη να δούμε τι αντίκτυπο έχουν όλα αυτά. Δεν είναι τώρα μαθηματική εξίσωση, δεν είναι δύο και δύο κάνουν τέσσερα Είναι μια βάση επί τη οποία χαράζεται πολιτική, η οποία πολιτική αποφασίζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λυπάμαι πάρα πολύ αν αυτό σας ενοχλεί. Δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά ήθελα απλώς να ξεκαθαρίσω ότι είναι μια πολύ συνειδητή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι μια απόφαση η οποία επάρθει εύκολα. Λύθει εύκολα. Ε, είχαμε διαφορετικές απόψεις και τελικά το Συλλογικό Όργανο των Επιτρόπων αποφάσισε πώς θα ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Α, είμαστε στην αρχή της διαδρομής και όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Είστε οι συνομοθέτες βεβαίως. Ευχαριστώ. Η κυρία Μανιάκη Γρίβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην ε, συνάδελφο η οποία έκανε την πρώτη αξιολόγηση και μπορεί καλύτερα να απαντήσει σε ερωτήσεις που έκαναν τα μέλη σας. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Άκουσα πολλές και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσες γίνεται. Καταρχήν, αν λείπουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Όχι, δεν νομίζω. Η κοινωνική εταίρη εκεί έγινε διαβούλευση στα πλαίσια της συμβουλευτική Επιτροπής για τα Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης σε μια ακρόαση του 13. Και η ΜΚΟ και αυτούς τους ακούσαμε το 15 σε μια ακρόαση. Βεβαίως η Διοικητική Επιτροπή για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό και βεβαίως την διαβουλευτήκαμε. Έγιναν και δύο διαβουλεύσεις διαδικτυακά, μία το 12-13 για το συντονισμό των μακροπρόθεσμων γονικών και επιδομάτων και επιδομάτων ανεργίας και έγινε άλλη μία το 15 για το συντονισμό των οικογενειακών επιδομάτων, του επιδόματος ανεργίας και επίσης ε, τους κανόνες για την απόσπαση. Οπότε για μένα η διαβούλευση έγινε. Δεν νομίζω πως έλειψε κάποιος. Για το κατά πόσο μας στήριξαν εμφανώς ή όχι οι ενδιαφερόμενοι, έχοντας διαβάσει εγώ την επιτροσιολογική μελέτη, καταλήγω στο εξής. Φαίνεται ξεκάθαρα πως η Διοικητική Επιτροπή έλαβε έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο και μας έδωσε πάρα πολύ τροφή και για, το, και για τα εναλλακτικά σενάρια, αλλά και παρουσίασε και δικά της εναλλακτικά σενάρια. Όμως καμιά φορά δεν ήταν απόλυτα εμφανής η συνεισφορά όλων. Τώρα για τη διασύνδεση με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και κατά πόσο αυτός ο σύνδεσμος λείπει. Αν κοιτάξετε τη μελέτη θα δείτε που στο παράρτημα 20, δηλαδή κοντά στο τέλος ενό πραγματικά μακροσκελούς εγγράφου, έχουμε δύο σελίδες, παράρτημα 20 για τις τεχνικές τοπολογίε για τις αποσπάσεις και θεωρώ πως δεδομένη δεδομένε σημασίας του θέματος θα ήταν πραγματικά χρήσιμο εάν κάποιες από αυτές τις πληροφορίες για τις αποσπάσεις και για το πώς συνδέονται με τα όσα ε, παρακολουθούμε είχαν τοποθετηθεί σε κάποιο πιο εμφανές σημείο της μελέτης μας. Επίσης, είχαμε την αιτιολογημένη γνώμη της γαλλικής γερουσίας και αυτό το οποίο μας είπαν το εξής κοίταξε το κατά πόσο ε, παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας γιατί οι εφαρμοστικέ πράξεις σύμφωνα με τις οποίες οι διαδικασίες θα ορισθούν από την Κομισιόν για το φορητό έγγραφο, ε, το αποδεκτικό το οποίο θα φέρει ο δικαιούχος κοινωνικής ασφάλισης δεν πέρασε από τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτή ήταν ουσιαστικά η γνωμοδότηση της Γαλλικής Γερουσίας.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 μου ζήτησαν ήδη οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου ε, ε, Μα με οι ερωτήσει που έκαναν, συμφωνώ με τι ερωτήσει που έκαναν και θα ήθελα να κάνω και μερικά σχόλια. Ε, ουσιαστικά μιλάμε για οικονομικά ανενεργούς πολίτες. Αυτό δεν είναι αρκετό όμως. Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη το ότι τα βασικά δικαιώματα μπορούν να περιοριστούν ε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Δίνω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Μπάλλα. Έχετε τη δυνατότητα να σχολιάσετε. Euh, euh, euh, Πολλά έχω να πω για τι απαντήσει που δόθηκαν ε, ειδικότερα από όσου ε, έκαναν την έρευνα αυτή. Και πολλά ερωτηματικά τίθενται για τις παρατηρήσεις που ακούσαμε. Όσον αφορά τη δημιουργική αναπροσαρμογή προς τα πάνω προς τα κάτω, όσον αφορά ε, τα οικογενειακά επιδόματα. Ε, εδώ πιστεύω έχουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, το θέμα του, του επιπλέον διοικητικού κόστους πρέπει να αξιολογείται είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων, αλλά υπάρχει ένα σημαντικότερο στοιχείο. Είναι το θέμα της αρχής. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος έχει πληρώσει εισφορές, γιατί από ό,τι θυμάμαι οι παροχές δεν είναι δωρεές, δεν είναι τσάμπα χρήματα. Είναι κομμάτι της αμοιβή που έχει παρακρατηθεί. Αν αποφασίζουμε λοιπόν ξαφνικά ότι τα οικογενειακά επιδόματα θα είναι λιγότερα διότι ένα παιδί βρίσκεται σε άλλη χώρα όπου το επίπεδο διαβίωση είναι φθηνότερο και το πώς θα αξιολογούμε αυτό το χαμηλότερο επίπεδο διαβίωση είναι άλλο ερώτημα. Χαμηλώνουμε δηλαδή αυτό το ποσό. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι ε, που παρακρατήθηκε από την αμοιβή του εν λόγω ατόμου του αφαιρείται. Κάτι το οποίο είναι άδικο. Αν είναι λοιπόν να κάτσουμε να εξετάσουμε το θέμα της ε, αναπροσαρμογής, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τις εισφορές των ε, εργαζομένων σύμφωνα με τα ποσά τα οποία θα μπορούσαν να τους παρασχεθούν ως παροχές. Έτσι γίνονται τα πράγματα εξαιρετικά περίπλοκα. Οπότε από μια έχουμε το διοικητικό κόστος και από την άλλη έχουμε την αρχή. Δύο πράγματα πρέπει να διαχωρίσουμε και να τα εξετάσουμε ξεχωριστά. Για το ζήτημα τώρα που συζητήσαμε τήθηκε για τα έντυπα Α1. Ε, είναι σημαντικό. Εγώ φοβάμαι το εξή. Η Κομισιόν έχει δίκιο που προτείνει αυτό προτείνει και μάλιστα πιστεύω ότι πρέπει να το τραβήξει και περισσότερο όσον αφορά τον έλεγχο των εντύπων Α1. Αλλά ουσιαστικά αυτό που πρέπει να ρωτηθεί κανεί σήμερα είναι κατά πόσο αποτελεσματικά αυτά τα έντυπα σήμερα. Βρισκόμαστε στον ψηφιακό κόσμο πλέον και χρησιμοποιούμε έντυπα, έντυπα περίπλοκα σε διαφορετικέ γλώσσε. Πώ θέλετε οι επιθεωρήσει εργασία να βρουν άκρη. πώς ε, οι διάφορες υπηρεσίες ε, των διαφορών χωρών θα κάνουν τη δουλειά τους ε, σοβαρά. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα εναρμόνισης των πληροφοριών αυτών μέσω σύγχρονων εργαλείων ψηφιακών ώστε να είναι καλύτερος ο έλεγχος, πιο αποτελεσματικός, πιο διαφανής, με χαμηλότερο διοικητικό κόστος και να υπενθυμίσω στους φιλελεύθερους και συντηρητικούς φίλους γιατί κατά ξέρω ότι θα το προσέξω αυτό που θα πω, μικρότερο διοικητικό φόρτο, με μικρότερο διοικητικό φόρτο για τι επιχειρήσει. Οπότε πρέπει να διερευνήσουμε αυτή την οδό. Έχει γίνει γελία η κατάσταση αυτή με τα έντυπα Α1 τη παλαιοληθική εποχή πλέον. Thank you very much. Ευχαριστώ. Χρονοδιάγραμμα. Θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση της, του σχεδίου έκθεσης στις 20 και 21 Νοεμβρίου εδώ στην Επιτροπή. Προθεσμία καταβολής τροπολογιών θα είναι 29 Νοεμβρίου, εξέταση τροπολογιών τον Ιανουάριο του 2018, σκιώδης, Φεβρουάριο και Μάρτιο, προθεσμία για σχόλια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και έγκριση στην Επιτροπή μας προβλέπεται να γίνει τον Σοφορία, δηλαδή τον Απρίλιο. Είναι φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα αυτό, γιατί απομένουν να γίνουν πολλά πράγματα. Ωραία, λοιπόν, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Καταπολέμηση ανισοτήτων ω μοχλό για την τόνωση τη δημιουργία θέσεων εργασία και τη ανάπτυξη. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Χάβι Λόπεζ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πρώτο σχέδιο της έκθεσής μου. Που έχει τίτλο, όπως είπατε, καταπολέμηση των νοσοτητών ως μοχλός για τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης. Όπως γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια οι ανισότητες ε, παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο λόγο και ειδικότερα Έχουμε δει πολλές εξελίξεις και πολλές συζητήσεις στον επιστημονικό κόσμο για το τι επίπτωση έχουν οι ανισότητες. Η Πρόεδρος διακόπτει καλώντας τους απερχομένους να φεύγουν ήσυχα. Όπως είπαμε λοιπόν υπήρξαν πολλές συζητήσεις για πώς επηρεάζουν οι ανισότητες ε, την οικονομία και πολλές ε, πτυχές της κοινωνίας. Ειδικότερα λόγω της ε, σοβαρής ύφεση και των συνεπειών που είχε στην Ευρώπη όσον αφορά τον καταμερισμό του πλούτου, την κατανομή του πλούτου Όλα αυτά σε σχέση με τη μαζική ανεργία που καταγράφηκε σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Η έκθεση αυτή λοιπόν αποσκοπεί να συμπεριληφθεί, να συλληφθούν οι ανισότητες ως αρνητικός παράγοντας και να αναγνωριστεί η ανάγκη καταπολέμησης των ανισοτήτων. Να θυμίσουμε ότι επανειλημμένως η Ευρωπαϊκή Ένωση στον οδικό χάρτη για την κοινωνική οικονομία, για την καταπολέμηση της ενεργείας, της στόχιας, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2020, της Ατζέντας της Λισαβόνας και ταυτόχρονα και οι συνθήκες προβλέπουν σύγκληση μεταξύ των στόχων της Ένωσης και σύγκληση μεταξύ των χωρών και καταπολέμηση της στόχιας είναι ελελένδετοι παραγόντες για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Αλλά δεν απαραίτητο το ίδιο πράγμα. Με την έκθεση αυτή λοιπόν θέλουμε πρώτα απ' όλα να εντάξουμε στο θεματολόγια μας τις ανισότητες ε, με σκοπό να τις ε, καταπολεμήσουμε. Ε, κατά δεύτερον, θέλουμε να αναγνωριστούν οι επιπτώσεις των ανισοτήτων σε δύο τομείς κυρίως ε, σε θέματα ηθικά ε, επηρεάζουν επίσης όμως και τον οικονομικό τομέα, την ζήτηση ουσιαστικά, την εξέλιξη της ζήτησης. Πολλά εγγραφά, πολλές μελέτες ε, επικυρώνουν αυτή τη θέση. Την έχουμε αναφέρει και εδώ κατά τις διαβουλεύσεις μας με διάφορους εμπειρογνώμονες. Στη συνέχεια, επίσης, οι ανισότητες εκ των πραγμάτων καταστρέφουν την εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Όπως γνωρίζουμε, οι πιο ίσες ε, κοινωνίες ε, είναι και πιο σταθερές, ε, διότι υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη από τα διάφορα στοιχεία της κοινωνίας. Υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη από τους πολίτες προς τους θεσμούς. Εφόσον λοιπόν αναγνωριστούν αυτές οι δύο διαστάσεις της ανισότητας, ε, θέτουμε το στόχο της καταπολέμησης και φτιάχνουμε έναν οδικό χάρτη που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών που ήδη έχουν γίνει στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οπότε υπάρχουν τρεις διαστάσεις που θα αναφέρω τώρα εν συντομία πρώτον. Η βούληση ε, χάραξης κοινωνικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ήδη μια εκθέση αναφορά όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτή. Πρόθεση είναι ε, να δημιουργήσουμε ένα βελτιωμένο κοινωνικό περιβάλλον πανευρωπαϊκά, βελτιώντα τι συνθήκε εργασία και βάσει και των καινοτομιών, των νέων στοιχείων στην αγορά εργασία. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη διαστασία αυτή. Δεύτερον, Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για την ευρωπαϊκή διάσταση των κοινωνικών πολιτικών. Θέλουμε να εισάγουμε και ένα στοιχείο το οποίο έχουμε ακούσει επανειλημμένως στην Επιτροπή μας την τροποποίηση του συντονισμού των οικονομικών, δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εντάσσουμε όλο και περισσότερο την κοινωνική διάσταση, γιατί και η κοινωνική διάσταση κινείται παράλληλα. Ε, να γίνουν λοιπόν συστάσεις προς τα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλίζουν και αυτά μια πραγματική ευημερία. Ξέρουμε ότι τα σημερινά συστήματα δεν λαμβάνουν υπόψη τις κοινοτομίες που έχουν εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία εντός της ε, κοινωνίας. Όλα τα συστήματα αυτά είναι από το μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην έκθεση επίσης γίνεται και μια αναφορά στις πιο ευάλωτες, πιο εκτεθειμένες ε, ομάδες ε, που είναι περισσότερο πιθανό να ε, βιώσουν τις ανισότητες, δηλαδή άτομα με αναπηρίες, άτομα που υποφέρουν από την ανισότητα λόγω η παιδική φτώχεια, η ηλικιωμένη, η δυσκολία πρόσβαση στην αγορά των, νεότερων, των νεωτέρων και γίνεται και μια ιδιαίτερη αναφορά στις πλέον ευάλωτες ομάδες οι οποίες βιώνουν από πρώτο χέρι τις ανισότητες. Πιστεύω λοιπόν ότι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε καλά και θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο αυτό μέσα στι επόμενε εβδομάδε, διότι αυτό είναι σίγουρα εφικτό και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει, πλέον πολύ σημαντική σε δημόσιο επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει ένα σαφές καθαρό μήνυμα ε, για το πόσο αναγκαίο είναι να καταπολεμηθούν οι ανισότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώσα αναχώρησε, οπότε πάμε κατευθείαν στην κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ κύριε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Χρειαζόμαστε περισσότερη ισότητα και σύγκληση. Αυτό θα αποδειχθεί αποφελές για όλους μας. Είναι πολύ σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ανάπτυξη. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πρώτα απ' όλα με δυσκολεύουν ε, οι άτυπες συμβάσεις εργασίας που εξορισμού θεωρούνται ερνητικές. Οι πιο ελαστικές μορφές εργασίας μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες για κάποιες ομάδες ατόμων. Έτσι λοιπόν ε, τα άτομα αυτά μπορούν να αποκτήσουν μια πρώτη ευκαιρία στην αγορά εργασίας έτσι μπορούμε να επανεντάξουμε στην αγορά στους του μακροχρονιά ανέργου, του συχνά ξεχνάμε. Δεύτερο μικρό πρόβλημα, η έκκληση για εξευρωπαϊσμό. Ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν ευρύτερη κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων και εναρμόνιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος για τους ανέργους, ε, μιας οδηγίας ε, για τις ε, μακροχρόνιες φροντίδες, ε, τις άδειες και τις συνθήκες εργασίας. Θα μπορούσα να σας στείλω ο σχετικό κατάλογο. Ε, πολλές ιδέες δεν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας ε, εδώ σε αυτήν την έκθεση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εφαρμόσουμε καταστολή στα κράτη-μέλη, να τα καταπιέσουμε. Πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές που είναι οι κατάλληλες για τους πολίτες τους οι ενιαίες λύσεις, το one size fits all, οι ενιαίες λύσεις για όλες τις περιπτώσεις τελικά μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά για κανέναν. Τρίτο, θα ήθελα να εκφράσω μια επιφύλαξη όσον αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Ας προσέξουμε στο αυτό που μας λέει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βελτιώσουμε την πρωτοβουλία. Τέλος, ε, θα ήθελα να πω ότι στην έκθεση ε, εντοπίζονται διάφορα προβλήματα ε, και απαιτούνται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, θα έπρεπε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τι λύσεις υπάρχουν ήδη για την τόνωση της αναπτυξής και της απασχόλησης και για να ευνοηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα. Ας υπογραμμίσουμε τον πυρήνα της έκθεσης αυτής και είμαι έτοιμη να, εργαστώ, και να συνεργαστώ επικοδομητικά με τον εισηγητή και τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Καλφασοβού. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω τα εξής. Να σας πω πως επιτέλους, επιτέλους γιατί περιμένω το θέμα αυτό να το συζητήσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και νομίζω ότι ήδη αυτό έχει αναγνωριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συγχαρώ το φίλο και συνάδελφο Χαβιέρ Λόπες γιατί Ε, ξεκίνησε αναλαμβάνοντας το βασικό κίνδυνο με αυτό το βασικό ε, κείμενο σε μια περιπέτεια ή πρόκληση ή ε, ελεύθερη πτώση δύσκολη και για το θέμα αυτό θέλω για, την, για το κουράγιο του θέλω να τον συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω. Τώρα, πρέπει να ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς σας τον τίτλο τον τίτλο που είναι «Η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην ως μοχλό για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης». Όταν ξεκινήσαμε να υπερασπιζόμαστε την ιδέα αυτή, στην ομάδα, η προσέγγιση που ακολουθούσαμε ήταν κάπως διαφορετική. Η γενικότερη ε, προσέγγιση ήταν διαφορετική από αυτή που ακολουθεί σήμερα ο εισηγητή μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες. Δεν θα θέλαμε αυτό τελικά να μας οδηγήσει στο να καταλήξουμε σε επιπτώσεις κοινωνικές οι οποίες θα προκαλέσουν διέρεση στο Κοινοβούλιο και όπου δεν είναι ε, σαφείς οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι πώς μπορούμε αυτή τη δυναμική της ανισότητας που είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ, γιατί δεν νομίζω ότι κανεί από εμά αισθάνεται ικανοποιημένο, πώ μπορούν αυτέ οι ανισότητε να φρενάρουν τη δημιουργία απασχόληση. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Πιστεύω, και στο σημείο αυτό θα επιμείνω, πως το διαστοτικό πρόβλημα με τις ανισότητες δεν ε, εξαρτώνται από το ε, τι γίνεται στο εξωτερικό, γιατί πρέπει να σου πω πως η κοινωνική πολιτική έχει ως σκοπό έχει ως σκοπό να ξεπεραστούν αυτές οι κοινωνικές ανισότητες και νομίζω ότι αυτό ξεπερνά κατά πολύ το πεδίο και των όσων εδώ θεσπίζουμε και των όσων έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Τι θα μειώσει τελικά την ανισότητα. Η αναδιανομητική πολιτική. Αυτό και μόνο. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της φορολογικής πολιτικής που θα ακολουθήσουμε. Γιατί μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού δεν νομίζω ότι πρόκειται να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Ούτε μέσω της εμπορικής πολιτικής. Νομίζω ότι είναι η βιομηχανική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, όλα αυτά τα οποία διαρθρώνουν μέσα στο πλαίσιο στο οποίο περιγράφουμε, που είναι η ανάπτυξη. Και στο σημείο αυτό μου λείπουν πολλά στοιχεία. Ε, Μπορώ βέβαια να σας παρουσιάσω ε, κάποιες από αυτές. Το κατόφλι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, το οποίο ομάδα μου θεωρεί πως θα έπρεπε να αποτελεί και εκτιμένο δικαίωμα. Νομίζω πως αυτό είναι ένα κατάλληλο μέτρο για να καταπολεμήσει τις ατομικές ε, ανισότητες, γιατί δημιουργεί ένα κατόφλι. Και αυτό μέσω των ισοδηματικών πολιτικών που εφαρμόζουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Οπότε το κατόφλι αυτό θα έπρεπε να μπει στον κοινωνικό πυλώνα και νομίζω ότι δεν βρίσκεται στον απόλυτο πυρήνα του κεκτημένου, αλλά είναι ο κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυναμική που δημιουργεί ανισότητε. Και μετά από αυτό πρέπει να προσθέσω μία σειρά από άλλε δράσει. Για παράδειγμα, η αγορά εργασία. Πώ ε, συνεισφέρει ή όχι στην ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αν κάποιος πιστεύει πως η ε, ανέλικτη αγορά εργασίας ε, επιτρέπει στο να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει την τελευταία έκθεση του ΩΣΑ που λέει όσο πιο μεγαλύτερη έλλειψη ευελιξίας έχει αγορά εργασίας, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ανεργία. Γιατί? Γιατί τότε οι επιχειρήσεις προχωρούν σε μετεγκατάσταση σε άλλες περιοχές όταν οι εργασίες τους είναι έντασης κεφαλαίων ή έντασης εργασιών. Οπότε πριν ξεκινούμε με τέτοιου είδου διεκδικήσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν οδηγούν πουθενά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν και κατόπιν τις βασικές κοινωνικές ιδέες, δηλαδή ομάδες που μειονεκτούν, θα ασχοληθούμε ή όχι. Είναι μια ανισότητα, η οποία από πού προκύπτει από την κακοτυχία, από την ίδια τη φύση, ε, από τις... γιατί μιλάμε και για αναπηρίες πολλές φορές. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ε, θα γίνονται εκεί οι περισσότερες προσπάθειες και νομίζω ότι αυτό δεν συνδυάζεται τόσο πολύ και καλό είναι που αναφέρεται εδώ, αλλά δεν έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα σπάσουμε τη δυναμική της ανισότητας και θα δημιουργήσουμε ε, απασχόληση. Γιατί? Γιατί αυτή η δυναμική καταστρέφει την ανάπτυξη και την απασχόληση, γιατί, γιατί δίνει χρηματοδότηση στο να ε, ελαφρύνει τις αρνητικές συνέπειες, αλλά δεν είναι αρκετό το να προχωρούμε σε μια τέτοια παρηγορητική τακτική. Πρέπει να σπάσουμε ε, όλη αυτή τη δυναμική. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε να διατηρείται αυτή η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ της αμοιβή, ε, αν κάνουμε δε τη σύγκριση μεταξύ κεφαλαίου και ε, εργαζομένου, γιατί έχουμε τα πάγια στο κεφάλαιο ε, και τα λοιπά τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε. Και θα κλείσω με αυτό στο οποίο ε, θα αναφερθώ τώρα κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να εξευρωπαίσουμε και αυτά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τους συντελεστές που αποδεικνύουν που εμείς μειώνουμε τη δυναμική της ανισότητας. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάτρικ Λεϊαρίκ δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει κανεί άλλο εδώ από την ΚΟΥΕ. Η Μόνικα Βάνα από του πράσινου. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Λόπε ε, για το σχέδιο έκθεση. Συμφωνώ μαζί σα απόλυτα όταν λέτε ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση από μόνη τη. Είναι πολύ σημαντική πιστεύω αυτή η έκθεση, όχι μόνο για αυτή την Επιτροπή αλλά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά την υποστηρίζουμε, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε κάποια κομμάτια και να συμπληρώσουμε κάποια που λείπουν. Χαίρομαι που αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανεργίας. Ε, ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα από τον Επίτροπο Άντορ για το Ευρωπαϊκό Επίδομα Ανεργίας. Ε, χαίρομαι που το ξαναθέτετε, αλλά λείπει κάτι πιστεύω. Τα πρότυπα για τους ανέργους ή για τους υποαπασχολουμένους δεν πρέπει να έχουν απλά μία μορφή σταθεροποιητή. Χρειαζόμαστε ελάχιστα κοινωνικά στάνταρ στην Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα, ε, ε, για τους ανέργους αλλά και υπό την ε, μορφή ενός συστήματος ελάχιστου εισοδήματος. Ως αντιστάθμισμα της ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης χρειαζόμαστε μια κοινωνική ένωση με συγκεκριμένα βήματα ώστε όχι απλά να έχουμε μια πιο κοινωνική Ευρώπη, όπως λέμε, ένα κοινωνικό πυλώνα, χρειαζόμαστε μια κοινωνική ένωση. Τα ελάχιστα πρότυπα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω, είναι απαραίτητα για εργαζομένους, για τους πιο ευάλωτους. Είναι σημαντικό ζήτημα. Εμείς θα, κάνουμε, θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ε, τίθεται θέμα αναδιανομής, αναδιανομής του πλούτου, των χρημάτων, των ευκαιριών. Και αυτό λείπει. Ε, και επίσης λείπει και η διάσταση του φύλου. Εκεί που μιλάτε για φτώχεια και καταπολέμηση της φτώχειας ε, και του κοινωνικού αποκλεισμού, προς το παρόν αναφέρεστε μόνο σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Είναι φυσικά πολύ σημαντικέ κατηγορίες και καλωσορίζουμε τις προτάσεις σας ε, στο κεφάλαιο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες στόχοι, για να τις πούμε έτσι, με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε. Του φίλου, τη διαστήση του φίλου, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και άλλες ομάδες στόχους. Επίσης θα θέλαμε να αναφέρεται στην έκθεση και ο ρόλος της ε, κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ. Όχι μόνο οι κοινωνικοί εταίροι και ε, τα συνδικάτα, ναι, παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά και η κοινωνία των πολιτών παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες ε, όσον αφορά την εξατομήκευση των φορολογικών συστημάτων και αυτό είναι σημαντικό. Το θέμα ουσιαστικά είναι επενδύσεις σε τελική ανάλυση. Εδώ λείπουν συγκεκριμένες προτάσεις από την έκθεση για το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις κοινωνικές επενδύσεις. Αναφέρεται για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που του λείπει μια κοινωνική υποδόμη. Μόνο το 5% του προϋπολογισμού του ΕΦΣΥ πάει σε κοινωνικές υποδομές. Αυτό είναι πρόβλημα, πρέπει να το αναφέρουμε. Και χρειαζόμαστε επενδύσεις για νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς, αξιοπρεπείς όχι απλά δουλειές, και χρειαζόμαστε και επενδύσεις σε πράσινες θέσεις εργασίας, στον τομέα της φροντίδας, της κοινωνικής ε, ασφάλισης, της εκπαίδευσης, ε, της κοινωνικής οικονομίας. Εδώ υπάρχουν αρκετές δυνατότητες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, και να εκφράσουμε πιο ρητά στην έκθεση αυτή. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελαστικότητα για τις χώρες που επιθυμούν να εφαρμόσουν ε, δημοσιονομική ε, εξυγίανση. Και η μακροοικονομική αιρεσιμότητα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Θα υποβάλουμε τροπολογίες, αλλά θεωρούμε ότι ήδη η έκθεση φυσικά αποτελεί μια εξαιρετική βάση. Ευχαριστούμε. Η Λαούρα Τζε δεν είναι εδώ, ο Μαραμπιτζότο. Ευχαριστώ λοιπόν για να αντισταθμίσουμε λίγο την πολυλογία του κυρίου Σαμπών. Θα ήθελα να ε, ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Μπιτζότο για την απουσία της. Ναι, έχουμε αρκετό χρόνο σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κάτι που δεν συνηθίζεται. Λοιπόν, να δω λίγο. Ο κύριος Γκουτιέρης έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χάβι Λόπες για αυτήν την πολύ σημαντική έκθεσή του. Είναι η πρώτη έκθεση που αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανισότητας ως οριζόντιο θέμα. Αναφέρονται οι αιτίες, οι επιπτώσεις, καθώς και μέτρα για να κλείσει αυτό το χάσμα που έχει ανοίξει στις κοινωνίες μας τα τελευταία χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, ε, οι ανισότητες οφείλονται σε τρεις αιτίες. Πρώτον, η κατανομή του πλούτου είναι άδικη και άνηση. Και νομίζω ότι με αυτή την άποψη συμφωνούν και πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο. Και κυρίως το θέμα της συγκέντρωσης των ε, κερδών που μετά δεν έκανε μια δίκαιη διανομή αυτών ε, υπέρ της ε, μέσης τάξης της μεσαίας τάξης ή των εργαζομένων, έχουμε μια κακή διανομή του πλούτου μέσω των μισθών και τα τελευταία χρόνια ως επίπτωση των πολιτικών λιτότητας που έχουν επιβληθεί στα, στις προνοιακές ε, διαδικασίες και το γεγονός πως ε, έχουμε μεγαλύτερη άμεση φορολόγηση και περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις, ε, μία αναδιανομή. Ε, οπότε νομίζω ότι όλα αυτά μας οδήγησαν στο σήμερα να έχουμε κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια βαθιά έλλειψη ανισότητας πάρα πολύ ανισότητα επίση σε επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματο, κάτι το οποίο πλήττει τη μεγάλη πλειοψηφία των ε, εργαζομένων. Και νομίζω ότι ο Χάβι Λόπες στην έκθεσή του περιγράφει ακριβώς αυτά τα προβλήματα και τις ελλείψεις ε, που έχουν τα δημοκρατικά μας συστήματα, όπως επίσης και τα κόμματα τα οποία με το μαγικό ραβδί λύνουν όλα τα προβλήματα και τα οποία θεωρούν πως ε, η ανισότητα είναι θέμα οικονομικό ή κοινωνικό για το οποίο φταίει μια συγκεκριμένη μερίδα του ε, πληθυσμού. Τέλος πάντων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί οι λύσεις που προτείνονται είναι μια κοινωνία η οποία θα ανακτήσει ε, την ε, ισότητα, η οποία θα μειώσει τις διαφορές και τις ανισότητες και η οποία θα ορίσει ένα καινούριο κοινωνικό σύμφωνο που θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Και όπως είπε ο, ο συνάδελφος θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές, τη βιομηχανική, την ενεργειακή, την ε, εμπορική. Ε, την κοινωνική έτσι ώστε να έχουμε ένα ελάχιστο ε, εγγυημένο εισόδημα έτσι ώστε να καταφέρουμε να βρούμε έναν νέο τρόπο φορολόγησης πραγματικά αναδιανεμητικής. Αυτό θα ήθελα να δούμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να αποδώσουμε τη δέουσα σημασία σε αυτή την έκθεση έτσι ώστε να ε, επαναπροσδιορίσουμε μια νέα κοινωνία με μια δίκαιη λύση έτσι ώστε να ξεφύγουμε όλοι από την κρίση. Τότε στην περίπτωση αυτή θα έχουμε εξυπηρετήσει και την κοινωνία ε, του μέλλοντος και τον ε, φιλοευρωπαϊσμό. Ευχαριστώ λοιπόν για μια φορά ακόμα το Βεχάβη για την καταπληκτική του δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Ριμπέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως ασαφή σε αυτή την έκθεση. Ποιο είναι το θέμα της έκθεσης τελικά. Καταπολέμηση των ανισοτήτων για να επιτύχουμε τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Αυτό ως αυτό, αυτός σκοπός ή σημαντικότερο κρίνεται η καταπολέμηση των ανισοτήτων. Ή αφετέρου θέλουμε να μιλήσουμε για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ε, οι, οι πολίτες να βρουν δουλειά. Γιατί αν το δούμε έτσι συγκεκριμένα το θέμα, είναι προφανές ότι θα αναγκαζόμασταν να κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν θέλουμε να επικεντρωθούμε στα ριζικά αίτια που αποτρέπουν ανθρώπους από το να βρουν δουλειά. κάποιος που ζει σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή, στις Αζόρες για παράδειγμα, τι εμπόδια αντιμετωπίζει. Ε, το ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο θέμα η παιδεία, η κατάρτιση. Πόσοι και πόσο δύσκολα βρίσκουν ε, μια θέση σε ε, ιδρύματα εκπαιδευτικά υψηλής ποιότητας. Γιατί αν δεν εξετάσουμε και αυτά τα ζητήματα, τότε στην ουσία αερολογούμε και καταλήγουμε σε μια έκθεση κενή περιεχομένου. Γι' αυτό και θα ήθελα να καλέσω τον εισηγητή να επικεντρωθεί στα ουσιώδη θέματα. Φυσικά η έκθεση, εντάξει θα μπορούσε κανείς να, να, την, ε, να την χαρακτηρίσει έως και ευχάριστη. Σημαντικό όμως αυτό που, που κρίνεται εδώ είναι να είμαστε συγκεκριμένοι. Ποιο είναι ακριβώς το θέμα της έκθεσης. Thank you, Madam. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. και όσα έχει ε, περιγράψει η ο οποίος πραγματικά είναι άξιος συγχαρητηρίων για τα όσα προσπαθεί εδώ να βάλει στην έκθεση και για τον τρόπο με τον οποίο θα μας βοηθήσει να πετύχουμε αυτά τα οποία επιθυμούμε. Όταν μιλάμε για ανισότητες και για τους λόγους που προέκυψαν αυτές οι ανισότητες, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στις βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως με αυτό που ε, περιγράφεται ως το έλλειμμα επενδύσεων, το οποίο προέκυψε από στη μετά την κρίση του 2008 ε, εποχή. Δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερβολικά ε, ασαφείς για το από πού πηγάζουν αυτές οι ανισότητες και πώς θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Νομίζω πως ε, αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια και των προσπαθειών για αύξηση της ανάπτυξης και της ανεργίας. Οπότε το πρώτο κομμάτι από το κύριο σώμα της έκθεσης όπου μιλά για συντονισμό ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανισότητας, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να εξετάσουμε πώς θα εξελίξουμε αυτές τις έννοιες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, με τον συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής και με όλα αυτά τα θέματα τα οποία καλύπτουν μία σειρά από κλάδους και που βέβαια θα οριοθετήσουν και το χώρο και τον τρόπο με τον οποίο θα προοδεύσει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω είχαμε μια ακρόαση εδώ χθες για τις ε, ε, μακροπρόθεσμες ε, ε, προοπτικές, ε, χρηματοδοτικές προοπτικές για την μετά το 2020 εποχή μιλήσαμε για την επίγουσα ανάγκη που υπάρχει να δούμε πώς αυτές λαμβάνουν υπόψη και το Brexit και την έλλειψη των 10 δις συνεισφοράς, όπως επίσης και τις επιπρόσθετες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν που έχουν να κάνουν με την άμυνα, με τη μετανάστευση, που χρειάζονται επιπλέον πόρους. Οπότε το κεντρικό σημείο είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα έλεγα πως η προστιθέμενη αξία εδώ είναι στη μείωση των ε, ε, ανισοτήτων. Δηλαδή, να ξεπεράσουμε το έλλειμμα επενδύσεων εκεί που είναι πιο τραγικό, μιλάμε για περιοχές στην Βουλγαρία που έχουν ΑΕΠ 10.000 ευρώ ε, κατ' Ε, και αυτό σε σύγκριση με περιοχές Γερμανία Γερμανίας που έχουν αντίστοιχο ΑΕΠ 60-70 Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια απερίφραστη ανισότητα. Και την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε μια έκθεση στο Στρασβούργο γιατί αυτή τη στιγμή ε, έχουν στα πλαίσια του ΕΦΣΙ ε, συμβασιοποιηθεί 91% των έργων στις, στα 15 κράτη-μέλη και 13% των επενδύσεων, και, συγγνώμη, και στο 10% για τα υπόλοιπα 13 κράτη-μέλη, τα οποία ξέρετε ποια είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε απολύτω σαφεί και να δούμε πώς μπορούμε να μπούμε στην πραγματική ουσία της συζήτησης ε, και να προχωρήσουμε στη συζήτηση αυτή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κύριε Χαβιλόπε, να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ε, ευρωβουλευτές, τους ε, σκιώδεις για όλα τα σχόλια που κάνανε. Σίγουρα θα μας βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερη δουλειά τις επόμενες εβδομάδες μέσω, ε, μέσω των τροπολογιών μας και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Αυτό που θα ήθελα είναι να κάνω ένα μικρό σχόλιο γενικότερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καταγράψουμε ε, τις δικές σας ε, παρατηρήσεις και θα ήθελα να πω το εξής. Για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η συνάδελφος κυρία Στίβενς μίλησε για το τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο και κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια εξατομίκευση των πολιτικών. Συμφωνώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε σκοπό εμείς να κόψουμε κουστούμάκι κατά παραγγελία για κανέναν. Υπάρχουν κάποια από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και προηγουμένως, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να έχουμε ένα κατόφλι για παράδειγμα ένα κοινό παρανομαστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και πέρα το κάθε κράτο μπορεί από εκεί και πάνω να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελεί και ένωση δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν κάποιες από τις νομοθεσίες που αυτή τη στιγμή γίνονται υπό, είναι υπό σήμερα, για παράδειγμα άδειες, μητρότητες και του και του, όπως συζητήθηκε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι του διαπραγματευσή αυτή τη στιγμή είναι ε, η επικουρικότητα μεν, αλλά και η ευρωπαϊκή διάσταση σε θέματα στα οποία μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες. Επίσης έγινε μια αναφορά στην αγορά εργασίας και αυτό από διάφορους συναδέλφους. Σίγουρα η ευελιξία στην αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνδέεται απαραίτητα με την ανασότητα, αλλά είναι όντως αλήθεια πως αυτές οι μεταλλάξεις αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια και αυτή η κατάτμιση και η διέρεση σε μόνιμες και μη θέσεις στην αγορά εργασίας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό, έχει οδηγήσει σε μείωση μισθών, αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το καταγράψω. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο αδύναμη η μισθή. Και αυτό έχουν να κάνει πολλέ φορέ και με τι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, θα το ξανασυζητήσουμε. Και αυτό στη διαδικασία των τροπολογιών. Και στους συναδέλφους από τους πράσινους να πω πως υπάρχουν βελτιώσεις, ναι. Οι ιδέες σας, για παράδειγμα, για τις επενδύσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Κάλβης. Εδώ πρέπει να δούμε το θέμα της αναδιανομής, πώς μπορεί αυτή η αναδιανομή να είναι πιο δίκαιη για όλους, πιο ισορροπημένη. Καταγράφω λοιπόν αυτά τα σχόλια. Οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ σας ευχαριστώ πάρα πολύ comentarios, ¿no? tanto de Brinsky como de, de Sergio, y, de, luego se ha hecho también una, una, un, un comentario. Και το Σέρχιο έκανε ένα πολύ ωραίο σχόλιο για τη φύση της έκθεσης και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Να δούμε δηλαδή πώς θέλουμε να το προσεγγίσουμε. Το μόνο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο τίτλος. Και νομίζω ότι τον είχαμε συμφωνήσει κιόλα. Όλες οι πολιτικές ομάδες γιατί είναι οι συντονιστές οι οποίοι συμφώνησαν τον τίτλο αυτό. Οπότε, η καταπολέμηση των ανισοτήτων είναι μοχλός για την τόνωση δημιουργία δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, πώς θα καταπολεμήσουμε την ανισότητα και γιατί η ανισότητα είναι σημαντική ε, στην οικονομία στην προσφορά ευκαιριών. Αυτή, αυτό είναι η λογική την οποία θα ακολουθήσει η έκθεση. Σίγουρα οι τροπολογίε θα συνεισφέρουν ε, στη βελτίωση του κειμένου, είμαι σίγουρος, και θα καταλήξουμε με μια προσέγγιση η οποία θα είναι κατάλληλη. Είμαι όμως πολύ σύμφωνος με τα σχόλια τα οποία έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να επιτύχουμε. Δεν είναι μόνο πολιτικό το μήνυμα που θα στείλουμε. Θέλουμε να δούμε τι θα πετύχουμε μέσω αυτής της έκθεσης και νομίζω ότι η υπενθύμηση αυτή είναι χρήσιμη και κυρίως ε, αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε τις εργασίες μας Και αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να λάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπαρόνα από την Γενική Διεύθυνση Προσχόληση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ονομάζομαι Μανώλα Γκέρινγκα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε για αυτή την έκθεση την οποία καλωσορίζουμε. Οι ανισότητες ε, βρίσκονται πάλι πραγματι στο επίκεντρο των εργασιών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ο πρόσφατος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Πυλώνας ε, για τα κοινωνικά δικαιώματα διασφαλίζει ένα σύνολο αρχών για την καλή λειτουργία των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των αγορών. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων αποτελεί το πυρήνα όλων αυτών, τόσο όσον αφορά τα αποτελέσματα που θα φέρει για καλύτερα εισοδήματα, αλλά και για την προσφορά ίσων ευκαιριών. Υπερασπιζόμαστε κάποιες στιβαρές αρχές εκεί, τις ευκαιρίες, την ισότητα των φύλων, την ε, φροντίδα και την παιδεία των παιδιών, ε, τη μακροχρόνια φροντίδα. Τα αναφέρομαι ε, διότι αναφέρθηκαν και κατά τη συζήτηση. Φυσικά, ο κοινωνικός πυλώνας λαμβάνει υπόψη και την επικουρικότητα. Όλοι καλούνται να υλοποιήσουν τον πυλώνα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Το εξάμεινο επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2017 εστιάστηκε σε μεγάλο βαθμό στην μείωση των ανισοτήτων. Επισημαίνει επίσης και τη σπουδαιότητα του φορολογικού συστήματος για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, αλλά έριξε φως και σε άλλα επίπεδα πολιτικής όπως ε, τα συστήματα παιδείας, υγείας και κοινωνικής προστασίας και πολλές συστάσεις εκδόθηκαν φέτος σε, για παράδειγμα, 8 κράτη-μέλη όπου υπήρξε μια πρόταση οκτώ συστάσεων για την επάρκεια και την κάλυψη. Ε, πέραν αυτών θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι παρότι ο πυλώνας ε, δημιουργεί αρχές ε, σύγκλησης προς τα πάνω, συνεχίζονται οι εργασίες και στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για το ελάχιστο εισόδημα μέσω της δημιουργίας ε, σημείων αναφοράς ε, στο πεδίο αυτό, κάτι που θεωρούμε σημαντικό και φυσικά ο πίνακας βαθμολογίας ε, περιλαμβάνει, προτείνει διάφορους δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της οικονομικής και κοινωνικής απόδοσης, ώστε να βεβαιωθούμε ότι πράγματι μπορούμε να αντιληφθούμε πού έχει σημειωθεί πρόοδος. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνο διάγραμμα το βλέπετε μπροστά σας. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 5η Ιουλίου. Εξέταση των τροπολογιών 30 με 31 Αυγούστου ψηφοφορία στην ΕΜΠΛ 28 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο του 2017. Έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα. Ε, έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη και θα συνεχίσουμε στις 3 το μεσημέρι με τις ψηφοφορίες. Οπότε μην ξεχάσετε να φέρετε τις κάρτες σας ε, για την ψηφοφορία και ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα το πρωί.